Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη δυσκολία επαναρχίζουμε μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δύσκολο να ξυπνήσει κανείς το πρωί. Δύσκολο να ξεπαρκάρει. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε το έργο μας γέρος. Πρώτο θέμα στην ημέρησια διάταξη είναι η έγκριση τη ημέρησιας διάταξης ελήψη αντιρρήσεων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η μέρηση διάταξη χωρίς καμία τροποποίηση. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Πρόεδρου για τις συστάσεις των συντονιστών της 12ης Ιουλίου. Έχουν ε, διανεμηθεί ηλεκτρονικά οι συστάσεις των συντονιστών, εάν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις μπορούν να εγκριθούν. Και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Προσκαλώ όλους τους συναδέλφους να βάλουν τις κάρτες στην ε, θέση τους και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. Όλες οι, όλα τα τμήματα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 2. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αμ, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 4. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. πέντε πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Έχετε ψηφίσει όλοι. Απορρίπτεται. Τέταρτη και τελευταία, τελευταίο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία η, 9 εκπίπτει, τροπολογία 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ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 με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Δεκτή. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες του προϋπολογισμού ομαδών 50-57 με 50-58 υπέρ κατά αποχές δεκτές 61-04 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61-02 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60-96 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα ψηφίσουμε τώρα το 60-81 το 2 υπέρ κατά αποχές δεκτό 60, 65 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 60-82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 60-83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60-84 υπέρ κατά <clears throat> απορρίπτεται. 60-56 υπέρ κατά αποχές δεκτο 60.76 60-76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-80 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 61-06 αποσύρεται. 61 ε, κατα Κατά. Αποχές δεκτό. 61-13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 61-08 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 61-05 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 61-14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 6109 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτό. 6107 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6110 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6127 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61-23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-39 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ομαδών από το 60-63 και 60-64 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 60-85 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60-65 υπέρ, <coughs> κατά, αποχές δεκτό. 60-86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60-66 υπέρ, κατά αποχές δεκτό 60-67 υπέρ κατά αποχές δεκτό 60-87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60-68 υπέρ κατά αποχές δεκτό 60-88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60-70 <clears throat> είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60-89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-71 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 60-91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-75 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 60-92 υπέρ κατά αποχες απόποχέ δεκτών. 61-30 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 61-11 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 61-21 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 61-18 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 61-26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69, 19, 61, 20 αποσύρθηκαν. 61, 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61, 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-40 υπέρ κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται Περνάμε στο 4 από κοινού την 60-73-74-99 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 60-90 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60-93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, από κοινού την 51, 52, 53 και 95 από κοινού τέσσερις μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. Από κοινού 59, 60, 61, 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε πάλι μαζί την 03, την 00, 01 και 98. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ομαδών πάλι την 77 με την 78 με την 79 με την 97. <clears throat> ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτές. Τώρα Adesso abbiamo un eh, emendamento orale. Τώρα έχουμε μια προφορική τροπολογία που θα σας παρουσιάσω σύντομα σχετικά με τα οργανογράμματα των εξωτερικών υπηρεσιών. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού. Οι υπηρεσίες αυτές βέβαια έχουν όλο και περισσότερες υποχρεώσεις λειτουργικού τύπου, καθήκοντα επιπλέον, τα οποία, οι οποίες ε, πίπτουν στις ε, υπηρεσίες αυτές και πολλές φορές οι εξωτερικοί πόροι είναι αυτοί οι οποίοι ε, καλύπτουν το κόστος των εργασιών, των δραστηριοτήτων που απευθύνονται προς τα έξω. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει μία τροπολογία για τη διατήρηση του οργανογράμματος των εξωτερικών υπηρεσιών. Αν είναι τέσσερις συνάδελφοι κατά της προφορικής, δεν τη θέτω σε ψηφοφορία. Είναι κάποιος κατά? Όχι. Καλώς λοιπόν. Τότε τη θέτουμε ε, συνολικά σε ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτές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 Συγγνώμη, πριν ξέχασα να κάνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Επανέρχομαι στο σημείο 3 της ημέρησης διάταξης. Όταν γύρισα τη σελίδα, πέρασα τις ανακοινώσεις και τις ξέχασα. Πριν περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης για τον ΕΚΑΟ, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, κάνω ένα βήμα πίσω για να σας ανακοινώσω ότι θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της ΕΜΒΗ στο Στρασβούργο 12 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο, του Στρασβούργου 7 με 9. Εκεί θα έρθει ο Επίτροπος Αρίας Καρανιέτη για να μας παρουσιάσει το Ναγκριθέν πακέτο για το κλίμα. Επίσης, ε, Δεδομένη της σημερινής ημερήσιας διάταξης, η απογευματινή συνεδρίαση 5η 29 Σεπτεμβρίου ε, θα πρέπει να παραμείνει. Δεν μας αρέσει και πολύ που είναι 5η απόγευμα, αλλά θα πρέπει να την κρατήσουμε και θα σας στείλουμε την ημερήσια διάταξη. Επίσης, η εξέταση τροπολογιών για την πρόταση για τα απόβλητα θα γίνει ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, στις 3 το απόγευμα, 5η απόγευμα, 29 Σεπτεμβρίου. Επίσης, να σας ανακοινώσω μια αλλαγή στη γραμματεία της Επιτροπής ΕΒΗ. Κυρία Χριστίνα Μάλμος ε, επέστρεψε στη γραμματεία της ΕΒΗ μετά από πολύχρονη θητεία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Σουηδικής Βουλής. Την ξανακαλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ, σηκωθείτε για να σας δουν όλοι, να δουν ποια είστε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Επιτροπή μας και πάλι. Επίσης, σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και ως συνήθως ε, σας έχουμε στείλει το φάκελο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-meeting και έχουμε και απευθείας αναμετάδοση της συνεδρίασής μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημέρης της διάταξης που αφορά το πρόγραμμα για το Παγκόσμιο Αγορακεντρικό Μέτρο της, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Ε, θα ενημερωθούμε για την έκβαση της συνεδρίας υψηλού επίπεδου πριν την συνέλευση της ΕΚΑΟ. Θα έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ, τον κύριο Χόλο Λέι, που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα υψηλού επίπεδου της ΕΚΑΟ. Παρακαλώ, κύριε Λέι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ επίσης τους ευρωβουλευτές που θα με ακούσουν και θα λάβουν μέρος στην ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί φέτος ε, θα γίνει η συνέλευση της ε, ΙΚΑΟ, του ΙΚΑΟ σε δύο εβδομάδες και εκεί δεν ε, μας παίρνει να αποτύχουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει όσο πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα και από περιβαλλοντική σκοπιά. Και εδώ έχουμε δύο σημεία αναφορά. Έχουμε τη Συμφωνία των Παρισίων και την απόφαση του ΔΟΠΑ, του ΙΚΑΟ, που έγινε πριν από τρία χρόνια στην προηγούμενη συνέλευση, με απόφαση να αναπτυχθεί ένα μηχανισμό, ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, GMBM, για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, για, ε, το, από το 2020, ώστε να αποφευθούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού ένα μέτρο όμως που θέλουμε να είναι ρεαλιστικό και εφικτό και να μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ε, ε, περιστάσεις, ε, τις διαφορετικές χωρητικότητες και να σεβαστούμε όλα τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Πάντως όλοι έχουμε επίγνωση του δύσκολου έργου που μας περιμένει, γιατί μερικές χώρες ε, δεν επιθυμούν τόσο φιλόδοξο αποτέλεσμα όπως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να, ε, να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Πάντως, αν επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ένα παγκόσμιο μηχανισμό για έναν οικονομικό κλάδο. Και είναι κάτι μοναδικό, πρωτοφανές και σίγουρα μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Θα πρέπει πάντως να τονίσω ότι στην ε, επερχόμενη συνέλευση του ΙΚΑΟ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις με πολλούς και διάφορους τρόπους και όχι μόνο με το παγκόσμιο Κεντρικό μέτρο του GMBM. Για παράδειγμα θα έχουμε στάνταρ για, τα, για τις εκπομπές του άνθρακα για τα νέα αεροσκάφη που θα εγκριθούν οι νέες προδιαγραφές και θα μας απαλλάξουν από 650 εκατομμύρια τόνους ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2040. Και από τη στιγμή που θα θεσπίσουμε τις νέες προδιαγραφές, σταδιακά θα τις κάνουμε και πιο αυστηρές. Κάτι που συνέβη και με το θόρυβο, τα επίπεδα θορύβου και τις εκπομπές ε, αζότου, τα οξύδια του αζότου. Επίσης, ε, στην προηγούμενη συνάδελφη, ο ΙΚΑΟ είχε αποφασίσει να καταλήξει μια δέσμη μέτρων ώστε να εξασφαλίσουμε το στόχο της βελτίωση ώστε να αναχαιτήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς. Αυτό προϋποθέτει κάποιες τεχνολογίες αεροναυπηγικής και βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα για την αεροπορία πέραν του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του GMBM. Οπότε το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο θα πρέπει να το εξετάσουμε μονομένα. Τώρα για τη διαδικασία. Πρόκειται για πολυσχηδείς διαπραγματεύσεις ε, και σίγουρα περίπλοκες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνη της. Ε, θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας στα πλαίσια του ΙΚΑΟ και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ και το επιτελείο του και εδώ και μήνες ε, ε, για να μην πω χρόνια, θα έχουμε έντονες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που τα μέλη της Επιτροπής σας ε, στη... έλαβαν μέρος στην ε, αποστολή υψηλού επίπεδου του προηγούμενου Μαΐου και χαίρομαι που θα λάβετε μέρος και στην συνέλευση του ΙΚΑΟ. Είναι σημαντικό οι βουλευτές να βλέπουν διεισόμαση την πορεία των διαπραγματεύσεων και και τον προηγούμενο Μάιο. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους ευρωβουλευτές που ήταν μέλη της αντιπροσωπείας. Ε, φυσικά εντείνονται οι διαπραγματεύσεις και την περασμένη εβδομάδα είχαμε τους φίλους του, της Προεδρίας στο Μόντρελ, καθώς ε, και την περασμένη Παρασκευή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ. Θα συνεχιστούν και συντονιστικές συνεδριάσεις, αυτή που θα γίνει στη Βρατισλάβα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και επίσης ε, είχαμε τις αντιπροσωπείες ε, στη συνέλευση της πολιτικής αεροπορίας. Εκεί ε, συμμετέχουν 44 ευρωπαϊκές χώρες που θέλουμε να συνταχθούν σε ένα κοινό στόχο. Και η Κορεπέρ θα συνεδράσει την επόμενη εβδομάδα και οι διμερείς επαφές με τις διάφορες χώρες θα συνεχιστούν εν ώψη της συνέλευσης που θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Τώρα για τα τεχνικά θέματα. Τα βασικά πολιτικά θέματα αποφασίζονται στην συνέλευση. Αλλά πρόκειται για ένα κινούμενο στόχο και η, συνέλευση, όπως γνωρίζετε, διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Και σε ό,τι αφορά το σχέδιο για την παρακολούθηση, υποβολή αναφορών και εξακρίβωση θα αρχίσει το 2019 και το Παγκόσμιο Αγοροκεντρικό Μέτρο θα αρχίσει σταδιακά από το 2021 να εφαρμόζεται. Η συμπερίληψη στο σχέδιο αυτό θα θα γίνει υποχρεωτική από το 2027 μέχρι το 2035 και η ειδική αναθεώρηση του 2032 θα κρίνει κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί ο μηχανισμός αυτός, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχουμε σε όλη τη δέσμη των μέτρων. Αυτά προς το παρόν αλλά όπω σα είπα, πρόκειται για μια εξελικτική διαδικασία για ένα κινούμενο στόχο. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, το σχέδιο απόφαση ε, περιέχει μια φάση οικειοθελού εισαγωγή ε, μέχρι το 2027 με ε, επιφύλαξη κάποιε εξαιρέσει. Πάντω, το Παγκόσμιο Κεντρικό Μέτρο, το GMBM, θεωρείται ω προκαταρκτική εναρκτήρια βάση πριν περάσουμε στην απαραίτητη μελλοντική υποχρεωτική φάση. είναι ένα σημαντικός τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε κοινέ αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες. Τώρα, η απόκληση των μικρών νησιωτικών χωρών, των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών με βάση τα ντεμίνιμις ε, λαμβάνεται υπόψη. Όλα τα κράτη, όσο μικρή πολιτική αεροπορία και να έχουν, ε, μπορούν εθελοντικά να ενταχθούν στο σύστημα. Πάντως εμείς θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι, όλες οι μείζονες χώρες ε, με μεγάλο κλάδο πολιτικής αεροπορίας να ενταχθούν από την αρχή στο σύστημα. Αυτό είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η φιλοδοξία μας και πιστεύω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στη συνεδρίαση που θα γίνει σήμερα και αύριο στην Πρατισλάβα ε, και θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο, ελπίζω να συμφωνήσουμε σε μια κοινή διακήρυξη ώστε και οι 44 χώρες του, της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της Πολιτικής Αεροπορίας να ενταχθούν από την αρχή στο σύστημα αυτό και το ίδιο και οι Ηνωμένε Πολιτείες ο Καναδά, ο Μεξικό και η Ινδονησία που ήδη έχουν υποσχεθεί ότι θα ενταχθούν από την αρχή στον μηχανισμό. Τώρα, τα βασικά μηνύματα. Θέλουμε ένα ε, παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο που θα είναι φιλόδοξο, ε, εύχριστο και με ευρεία συμμετοχή ήδη από την αρχή, όσο πιο ευρεία γίνεται. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θα δούμε όμως τι προσπάθειες θα καταβληθούν και από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Γιατί η παγκόσμια ανάπτυξη και η ανάπτυξη παγκόσμιας πολιτικής αεροπορίας μέχρι το 2020 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θέλουμε καλόπιστα να επιδιώξουμε πρόοδο και με τις υπόλοιπες χώρες, ακόμη και με τις αναπτυσσόμενες που αναπτύσσουμε ταχύς ρυθμούς την πολιτική τους αεροπορία και ε, τακτική έλεγχη και αναθεωρήσεις και αξιολογήσεις ε, θα κρίνουν το ύψος και των φιλοδοξιών μας και πρόθεσμα. Πάντως πιστεύαμε ανέκαθεν ότι η τακτική αναπηρετή έκθεση είναι απαραίτητη για να έχουμε ε, μια ανάπτυξη που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτό αναφέρεται και αντικαταπτυρίζεται και στο σχέδιο ψηφίσματος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα η συνέλευση δεν είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας συνεργασίας. Θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη σκληρή δουλειά για να εφαρμόσουμε ε, τα μέτρα που θα θεσπίσουμε. Και το σχέδιο ψηφίσματος για το Παγκόσμιο Αγοροκεντρικό Μέτρο θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα οδικό χάρτη για όλες τις εκκρεμότητες που θα πρέπει να διαθετηθούν ώστε να ξεκινήσει το MRE το 2019 και το Παγκόσμιο Αγοροκεντρικό Μέτρο το 2021. Κάτι που προϋποθέτει σκληρή δουλειά και μεγάλη προσήλωση στο σκοπό. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να λιάνουμε τα προβλήματα με την καταχώρηση, με τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εξακρίβωσης και στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών είχαμε μία πιλωτική φάση και μία προσέγγιση αναφάσης και σταδιακή ε, προβλέπεται και για το Παγκόσμιο Αγορακεντρικό Μέτρο. Διαφοροποιημένη αλλά υπεύθυνη θέση. Και μέχρι το 2027 η κάλυψη του μέτρου θα αυξηθεί Γι' αυτό θέλουμε να παροτρύνουμε όσο δυνατό περισσότερες χώρες να ενταχθούν στο μέτρο αυτό από την αρχή. Γιατί ο περιβαλλοντικός του αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των χωρών που θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο αυτό σε προώρη φάση. Πρέπει να περιμένουμε να γίνει συνέλευση του ΙΚΑΟ μέχρι να λάβουμε αποφάσει. Θα ήταν πρόωρο να κάνω δηλώσεις πριν από τη συνεδρίαση αυτή έχουμε συμφωνήσει να δώσουμε στον ΙΚΑΟ την ευκαιρία να επιτύχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την Επιτροπή είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτή τη συνέλευση. Καταληκτικά, η Επίτροπος Μπούλτ και εγώ και οι ε, αρμόδιοι τη DG Move και τη DG για την, ε, για την, κλιματική αλλαγή και εκπρόσωποι τη ΕΑΣΑ θα είναι παρόντες σε αυτή την διάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή υποστηρίζει ιδιαίτερα και περιμένει ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς στην διάσκεψη του ΙΚΑ. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι καλόδεκτα και θα είναι μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε και με τη συνάντηση υψηλού επίπεδου τον προηγούμενο Μάιο και είμαι στη διαθεσή σας για να ακούσω τις απόψεις και να απαντήσω ενδεχομένως σε ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Thank ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με την Γκέρλινγκ, μέλος της αντιπροσωπείας μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χολολάη για τη φροντίδα που έδειξε στο ταξίδι μας, εμάς κατά τη διάρκεια του ταξίδιου τον Μάιο ε, γενικά είχαμε μια δύσκολη αρχή όταν πήγαμε στη συνάντηση αυτή για πρώτη φορά το Φεβρουάριο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα όμως. Είχαμε διμερείς επαφές με άλλα μέλη του ΙΚΑΟ και ήταν ενδιαφέρον στη συνάντηση εκ νέου τον Μάιο να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα νιώσαμε τον Μάιο ότι ήμασταν τμήμα της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αντίληψης. Παρ' όλα αυτά έχουμε διαφορές μεταξύ μας, δεν το ξεχνάμε αυτό, και σαν κοινοβούλιο δεν είμαστε διαπραγματευτές, προσπαθούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα προς κάποιες κατευθύνσεις και είδαμε πολλά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΙΚΑΟ. Πάντα ακούμε για μυστικότητα και για έλλειψη διαφάνειας. Αυτή τη στιγμή όμως βρήκαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε ανοιχτά με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε οι διμερείς επαφές μας με τα άλλα μέλη του ΙΚΑΟ ήταν λίγο πιο επιφυλακτικές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με πολιτική αποστολή αλλά και διπλωματική αποστολή. Αυτό είναι δύσκολο για τους κοινοβουλευτικούς. Ξέρετε ότι έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και δεν έχουμε πάντα την δυνατότητα να εκφραστούμε με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε εδώ. Τώρα για τα θέματα που αφορούν την μυστικότητα κτλ θα πρέπει να σημειώσουμε την διαφορά που, που υπάρχει ανάμεσα στο πώς βλέπουμε εμείς τον μηχανισμό αυτό και στο πώς το βλέπει το ΙΚΑΟ. Αν πάρετε σαν παράδειγμα τη Συμφωνία των Παρισίων, εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική αεροπορία σήμερα ε, τις ε, χαρίστηκαν ουσιαστικά. Είναι ανεξήγητο ε, το πώς πήραν μια τέτοια εξαίρεση από τις υποχρεώσεις τους. Ενώ το ΙΚΑΟ πιστεύει ότι ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ περίεργο, απλά τους επένεσε η διεθνής κοινότητα γιατί πηγαίνουν καλά, κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Έχει σημασία λοιπόν Εμεί σαν μέλη που δεν εμπλεκόμεθα άμεσα με το θέμα αυτό να καταλαούμε τις απόψεις των άλλων. Και έρχομαι πάντα στο θέμα της μυστικότητας και θα θέσω και την ερώτησή μου. Οι φίλοι της Προεδρίας συναντήθηκαν εδώ και λίγες μέρες ε, και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά για την έκβαση αυτής της συνάντησης. Ε, ε, και κάποιες ε, αναφορές που γίνονται στο site της ΙΚΑΟ δεν δείχνουν τίποτα. Μπορεί ο κύριος Χολολάης να μας μπορέσει να μας προσανατολίσει λίγο σε σχέση με τη συνεδρίαση αυτής της ομάδας. Οι επαφές που έχω με δημοσιογράφους μου λέγουν ότι μια συμφωνία, βέβαια το ΙΚΑΟ δεν θα το πει ποτέ συμφωνία, αλλά μια κάποια συζήτηση που θα οδηγήσει σε συνένεση ε, δημιουργείται επί τη βάση αυτής της εθελοντικής προσπάθειας, όχι υποχρεωτικής. Ε, μπορεί να μας διαφωτίσει ο κύριος Χολολάης λοιπόν. Είπατε επίσης ότι ένα βασικό θέμα για μας είναι η διάσκεψη έτσι ώστε όλες οι χώρες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξ αρχής. Ε, έχουμε όμως και κάποια άλλα θέματα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή διαδικασία αναθεώρησης και να διασφαλίσουμε επίσης την αξιοπιστία και την πραγματική σημασία των ε, credits, των ε, που ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και να δούμε τι θα γίνει και με τη θέση των ΙΠΑ, η οποία συνδέεται με το ευρωπαϊκό ETS, γιατί εμείς είχαμε προτείνει ε, τα GMBM να λαμβάνουν υπόψη ε, και άλλα γεωγραφικά σχήματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Thank you very much. And now Mr. Gerbrandi. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ολολέη για τα λόγια του. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπε η Τζούλι Γκέρλινγκ. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά στην Επιτροπή αυτή. Αυτό καταδεικνύει την ενότητα της Επιτροπής μας για το ζήτημα αυτό. Έχω κάποια ερωτήματα προς την Κομισιόν και κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις επί τη βάση των τελευταίων εξελίξεων και επίσης μετά από την ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας πριν από λίγους μήνες. Η ΙΚΑΟ είχε δεσμευτεί να υπάρξει ουδέτερη σε σχέση με τις εκπομπές άνθρακα ανάπτυξη μετά από το 2020. Εμείς συμφωνήσαμε με αυτή τη δέσμευση. Αν δείτε όμως τώρα τα έγγραφά τους, απέχουν πόρο από το να είναι ουδέτερη σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος το 2020. Μόνο από το 2027 θα είναι υποχρεωτικό να γίνεται κάτι τέτοιο και ακόμα και τότε υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εξαιρεθούν κάποιες χώρες από αυτή την υποχρέωση. Εγώ κατάλαβα ότι επί βάση των <clears throat> ορισμών που είχαμε συμφωνήσει, ακόμα και χώρες όπως η Ιταλία και το Βέλιο δεν θα είχαν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτό το σχήμα. Δεν ανησυχώ για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί νομίζω θα προσχωρήσουν ως ομάδα. Αλλά τι μας λέει αυτό για τη γενική προσέγγιση όταν βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές δεν εμπίπτουν στους ορισμούς που θα τους υποχρεώσουν να προσχωρήσουν σε αυτό το σχήμα. Και μόνο από το 2027 θα είναι υποχρεωτική η προσχώρησή τους, 7 χρόνια μετά από την αρχική δέσμευση που είχε αναλάβει η ΚΑΟ. <coughs> Δεύτερον, και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο στο Μοντρεάλ, η ΙΑΤΑ, η Διεθνής <clears throat> Ένωση Πολιτικής Αεροπορίας, κάνα τους δικούς υπολογισμούς και μίλησαν για ένα οριακό κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες. <clears throat> Έτσι ξεπερνάμε την αρχική συζήτηση για το κόστος γίνεται πιο πολιτική η συζήτηση. Αν είναι οριακό το κόστος και επί τη βάση υπολογισμών αυτών που θα πρέπει να επομιστούν αυτό το κόστος, γιατί κάνουν τέτοια φασαρία οι πολιτικοί. Αυτό είναι πιο πολιτικού χαρακτήρα από την προηγούμενη συζήτηση για το κόστος. Και αυτό είναι και η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτών που είχαμε συμφωνήσει στη διάσκεψη των Παρισίων. Αν δούμε τα στοιχεία, την πορεία των διαπραγματεύσεων, νομίζω δεν κάνουμε πολλά πράγματα. Συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πόσο τμήμα της αύξησης της εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μετά από το 2020 θα καλυφθεί από τα μέτρα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα το Μάιο, 50% του συνόλου θα καλυφθεί από αυτό το σύστημα. Μα πώς μπορείτε να μιλάτε για ουδετερότητα σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος όταν καλύπτεται από το σύστημα αυτό μόνο το μισό των εκπομπών. Δεν έχει νόημα. Και επίσης η Ιουλία Γκέρλινγκ μίλησε για την ποιότητα των αντισταθμιστικών μέτρων. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται ότι μπόρεσε να το συζητήσει ο ΙΚΑΟ και αυτό δείχνει και πάλι τον ερμητικό χαρακτήρα <clears throat> των συζητήσεων του ΙΚΑΟ. Ο ΙΚΑΟ πιστεύει ότι αυτοί θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για την ποιότητα των αντισταθμίσεων. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται η αντιστάθμιση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, αλλά αυτοί θα πρέπει να κρίνουν αν είναι ικανοποιητικέ αυτέ οι αντισταθμίσει, Ίσως έχετε να μα πείτε κάτι γι' αυτό. Και το τελευταίο μου ερώτημα αφορά τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με περιφερειακά συστήματα για τις εκπομπές. Γιατί αυτό σε τελική ανάλυση είναι και το ουσιαστικό. Θέλουμε όλοι να έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία, αλλά τα συστήματα εμπορίας εκπομπών για διεθνείς πτήσεις δεν θέλουμε να τα χάσουμε και επομένως αν <clears throat> υπάρξει εξαίρεση των περιφερειακών πτήσεων από τον ΙΚΑ, αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα εκπομπών. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής χρειάζονται διεθνεί λύσης και οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν πάει στο Μοτρεάλ και θέλουν να προωθήσουν αυτήν την λύση θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο κτλ. σε μια τέτοια λύση. Εγώ χαίρομαι για το γεγονό ότι ο ίδιο ο αεροπορικό κλάδο έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο μέχρι το 2020 να μειωθούν κατά ίμιση οι εκπομπές. Και επειδή εμείς θέλουμε μια διεθνή λύση, εμείς έχουμε δύο φορές ε, εξαιρέσει την, τον αεροπορικό κλάδο από το ETS, από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αλλά αυτό το οποίο τώρα είναι σημαντικό είναι ότι η νομοθεσία που ισχύει τώρα, ακόμα και δεν την αλλάξουμε, η τωρινή νομοθεσία να έχει πλήρη εφαρμογή από του χρόνου. Και βάσει αυτής της νομοθεσίας θα εφαρμοστεί πλήρως αυτή η νομοθεσία σε διυπηρετικές πτήσεις που έρχονται ή φεύγουν από την Ευρώπη όταν υπάρξει μια πραγματική συμφωνία στον ΙΚΑΟ για τη μείωση των εκπομπών. Όπως είπε η κυρία Γκέρλιν και ο κύριος Χερ Μπράντι, αυτό το οποίο προτείνεται από τον ΙΚΑΟ δεν είναι πραγματική μείωση. Αυτό το οποίο λέει ο ΙΚΑΟ ως ανάπτυξη η οποία θα είναι η οποία θα είναι ουδέτερη σε σχέση με τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο, αυτό αφορά μονάχα την περαιτέρω ανάπτυξη. Επίση, το θέμα των αντισταθμίσεων, το θέμα τη ποιότητα των αντισταθμισμάτων δεν έχει ρυθμιστεί. Εμείς έχουμε μία νομοθετική πρόταση η οποία θα καταργήσει τα αντισταθμίσματα για άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Παραδείγματος χάρη, για τη χαλιβουργία. Λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει μόνο ο αεροπορικό κλάδο ο οποίο θα έχει αυτά τα αντισταθμίσματα, αν οι άλλοι κλάδοι δεν θα έχουν τίποτα. Ο εκπρόσωπο τη δική μου χώρα, τη Γερμανία, σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, εξέφρασε μια θέση η οποία ήταν προσωπική κατά κάποιο τρόπο, δεν ήταν θέση της κυβέρνησης, και ζήτησε να υπάρξει μια πιλωτική φάση. Αν δούμε όμως τη συνολική κατάσταση, όλα αυτά που έχουν γίνει μετά τη διάσκεψη των Παρισίων για τον αεροπορικό κλάδο, εμείς θέλουμε πάντα να είναι ο τομέας αυτός φιλόδοξος. Η χαλιβουργία έχει διαμαρτυρηθεί και, και δικαιολογημένα. Θα πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερο περιθώριο για ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να περιορίζεται μονάχα εκεί η φιλοδοξία για τη μείωση των εκπομπών. Αυτά λοιπόν τα οποία συζητά ο ΙΚΑΟ πρέπει να είναι φιλόδοξα. Το να μιλήσουμε τώρα σε μια πιλωτική φάση, εγώ <clears throat> πιστεύω ότι για την κλιματική αλλαγή δεν βρισκόμαστε πια στην εποχή των ασαφών συζητήσεων, των γενικών συζητήσεων υπάρχει μια σαφής και σοβαρή ε, υποχρέωση που έχει αναλάβει η διεθνής κοινότητα για να λυθεί το πρόβλημα των εκπομπών. Ο οποιοδήποτε λοιπόν είναι υπεύθυνο, η μηχανική, η, η αρμόδιοι στην, ε, στον αεροπορικό κλάδο δεν μπορούν να φέρουν κατά κάποιο τρόπο τον κλιματικό αεροσκάφος σε πορεία πτώσης. Είναι πολύ σοβαρό αν γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να είμαστε σε μια πειραματική φάση όπως ζητούν ορισμένοι για μια πιλωτική φάση. Θα πρέπει να δράσουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι αποφασιστικός. Για να είμαι συγκεκριμένος, με τρομάζει η ιδέα ότι είμαστε ακόμα για ορισμένους σε μια πιλωτική φάση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από το 2005 να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για μια πιλωτική φάση. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε μονάχα στα σπάργανα στις προσπάθειές μα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να απορρίψει μια διεθνή συμφωνία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό τις επόμενες εβδομάδες, να πετύχουμε κάποια διεθνή συμφωνία. Η οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη από την απουσία μιας συμφωνίας, αλλά υπάρχει και εδώ ένα σημαντικό σημείο αποφασιστικού χαρακτήρα αν αποφασιστεί στο Μοντρεάλ ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας σύστημα ETS για τον αεροπορικό κλάδο, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως το Κοινοβούλιο μας, η Επιτροπή μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο ισχνό αποτέλεσμα να διατηρηθεί το ETS μονάχα για τον αεροπορικό κλάδο μόνο μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει και μεγαλύτερη ισοδικία για άλλους βιομηχανικούς κλάδους όπως είναι η χαλιβουργία, εάν είμαστε τόσο επίκης για τον αεροπορικό κλάδο. Και αυτή τη στιγμή Ξέρουμε ότι ο ΙΚΑΟ δεν έχει αποφασίσει ουσιαστικά τι θα γίνει μέχρι το 2027. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω λοιπόν είναι αν η Κομισιόν ή τα κάτι μελη που θα διαπραγματευτούν στη Σύνοδο του ΙΚΑΟ στο Μαντρεάλ υπογράψουν μια συμφωνία η οποία ανατρέπει ουσιαστικά την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει τώρα, αυτό θα είναι σοβαρή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Και ελπίζω ότι έχει επίγνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία πρέπει να υπερασπιστούμε. Γι' αυτό το δικό μου πραγματικό ερώτημα είναι, είναι σαφές στην Κομισιόν και το έχετε τονίσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν επιδέχεται ερμηνείες ή όχι. Σας ευχαριστώ κύριε Σέικχοτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έδειξαν τέτοια ευγένεια και έτσι εγώ δεν χρειάζεται να είμαι τόσο διπλωματικός, γιατί οι εισαγωγικέ παρατηρήσεις ε, ε, με σόκαραν. Φαίνεται σαν να είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εκπρόσωπος του ΙΚΑΟ. Νόμιζα ότι ήσασταν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε υπάρχει μία δέσμη μέτρων. Αυτά μας λέει και ο ΙΚΑΟ κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Μόντρελ. Ότι θα έχουμε μελλοντικέ τεχνολογίες για τα βιοκαύσιμα, για τα αεροσκάφη που δεν είναι όμως για σήμερα αύριο. Μιλάμε ουσιαστικά για το απότερο μέλλον και επίση έχουμε προδιαγραφή διοξιδίου του άνθρακα. Πότε όμως θα τεθεί σε ισχύ? Από το 2027 και μετά. Οπότε τι να... δεν θα μας βοηθήσει καθόλου, δεν θα μας εξυπηρετήσει ούτε την επόμενη δεκαετία αλλά ούτε και μετά γιατί ε, το 90% των αεροπλάνων Airbus και, που είναι Airbus και Boeing δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αποδοτικότητας που έχετε. Ελπίζω να μην φτιάχνουμε αυτόν τον τρόπο και πολιτικές για τις κλιματικές αλλαγές. Ναι, υπάρχει δέσμη μέτρων, αλλά τι να πω. Δεν έχει τίποτα ουσιαστικό αυτή η δέσμη μέτρων. Και γι' αυτό για την Ευρώπη ένα παγκόσμιο τέτοιο μέτρο αγορακεντρικό, GMBM, ήταν πολύ σημαντικό μέτρο. Και από ό,τι θυμάμαι είχαμε πει ανέκαθεν στην Ευρώπη ότι το GMBM θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2021. Τελεία και παύλα. Τώρα ξαφνικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει είχαμε πιλωτική φάση και για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αυτό όμω έγινε πριν από 10 χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν ακόμη μιλούμε για πιλωτικές φάσεις και πειραματικές φάσεις, τι να πω. Είναι αυτή η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σα έκαναν πλήση εγκεφάλου στο Μόντρεαλ. Μην μας λέτε τέτοια πράγματα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το ETS. Η Κίνα έχει πιλωτικέ φάσει τώρα για το ETS. Μην μιλάμε για πειραματικέ φάσει που θα ξεκινήσουν μετά από μια πενταετία. Επίση, είπατε ότι ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει μια σταδιακή εισαγωγή. Τι μιλάμε όμω τώρα. Μιλάμε για ένα εθελοντικό σύστημα μέχρι το 2027 και από το 2027 και μετά πάρει, πάντα υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης που θα πρέπει να εξεταστεί στη συνέχεια με την κριτήρια θα ισχύσει. Οπότε η σταδιακή ένταξη θα ξεκινήσει τώρα και, το, και μιλάμε για ένα παγκόσμιο μέτρο GMBM που θα ξεκινήσει το 2027 και από εκεί θα ξεκινήσει μετά η σταδιακή ένταξη. Τεράστια διαφορά και απόκληση από την αρχική μας συμφωνία. Απαράδεκτο. Ποιο είναι το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται να υποκληθήκαμε ε, το Σεπτέμβριο στο Μόντριελ, στο Νικάο. Και πραγματικά αυτό είναι απαράδεκτο και πραγματικά είναι σαν να ξεπουλάμε όλες μας τις αρχές και τις αξίες. Εμείς θέλουμε ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, ένα παγκόσμιο GMDM που θα ξεκινάει το 2021. Δεν θέλουμε ούτε πιλωτικό, ούτε περιοματικό, ούτε θελοντικό σύστημα, αλλά είναι υποχρεωτικό που να ξεκινάει το 2021 και μπορεί να υπάρχει ίσως μια σταδιακή ένταξη κάποιων χωρών, αλλά με ποια κριτήρια θα πρέπει να τα ξέρουμε από τώρα. Αυτό να συζητήσουμε. Και ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήδη έχει συνθηκολογήσει και θα πάει στην Πρατισλάβα ή αλλού, ευελπιστώντας ότι θα πείσει και άλλες χώρες να ενταχθούν και ο θελός στο σύστημα αυτό που είναι θελοντικό, είναι προαιρετικό ούτως ή άλλως. Δεν ξεκινήσαμε από αυτό το σημείο αφετηρίας, αλλά τα λέγαμε. Βέβαια ο Πίτερ είναι πολύ ευγενικό. λέει να μην το μπλοκάρουμε. Εγώ δεν βλέπω λόγο να το εγκρίνουμε πάντω. Και αν επιπλέον δεν επιτρέπονται καν τα περιφερειακά συστήματα, τι να σα πω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ελπίζω να διατρανώσουμε τη γνώμη μας και να ε, υψώσουμε μια πιο ηχηρή φωνή και να είμαστε λίγο πιο, να δείξουμε μεγαλύτερη πυγμή από ό,τι σήμερα. Γιατί αυτά που τα λέμε, που ακούμε από το Μόντρεαλ, ελπίζω να είναι διαφορετικά, να μην ε, προσυπογράφουμε τη γραμμή του Μόντρεαλ και του ΙΚΑΟ. Ελπίζω να έχουμε δική μας θέση. Εκτός και αν μετά από μια πενταετία ε, προσληφθείτε στο Μόντρεαλ και αρχίσετε να δουλεύετε εκεί. Εμείς ως πολιτικοί κάποιες φορές χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε και σε άλλες ε, μορφές διπλωματίας, αλλά εγώ πραγματικά θα υψώσω τη φωνή μου στο Μόντρελ. Μπορεί να είμαι κάπως πιο διπλωματικός, ό,τι σήμερα και λιγότερο ε, ομός και απότομος, γιατί με επηρεάζει θετικά η Τζούλη, αλλά αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα, αυτό θα πω κυρίως, ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Η κυρία Σερ Πιέρικ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές, Πρόεδρε, ότι η συζήτηση που προηγήθηκε παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να ομολογήσω ότι και εγώ η ίδια έχω επηρεαστεί από αυτά τα οποία άκουσα από τον Ολλανδό συνάδελφο. Ξέρω ότι οι ανησυχίες είναι πάρα πολλές και για τις εκπομπές καυσαερίων αλλά και για την διατήρηση του τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Μιλήσαμε επίσης ε, για τη Γεωργία νωρίτερα. Ε, δεν ξεχνάμε ότι είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας για την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις να θέσω. Αναφερόμαστε στις πτήσεις ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο διεθνής. Ε, ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας ε, αποτελείται και από πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν την δραστηριότητά τους και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αγοράζουν έτσι δικαιώματα εκπομπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως από τους κανονισμούς της ΕΚΑΟ και μας λέγουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι κινδυνεύουν να χάσουν τμήματα των αγορών. Ε, θα λειτουργήσει δηλαδή η αναδιοργάνωση της αγοράς ε, προς όφελος του Ντουμπάι, προς όφελος της λαϊκής Κίνας και εις βάρος των αεροπορικών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη και μετά θα πάρει το λόγο η Επιτροπή για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ αγαπητά μέλη για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Για την ειλικρίνειά σας επίσης και την ευθύτητά σας. Κάτι το οποίο θα στηρίξει ακόμα περισσότερο τα επιχειρήματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Εμείς προσπαθούμε ε, στην Τραν να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να πετύχουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Όπως είπα, η, τα χρονοδιαγράσματα της λειτουργίας των μηχανισμών δεν είναι δεδομένα και πολύ θα θέλαμε ένας μηχανισμός να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το 2021. Από την άλλη όμως δεν είμαστε μόνοι μας και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος το ταχύτερο δυνατόν με υποχρεωτικό τρόπο. Υπάρχουν όμως και άλλοι εταίροι στη διεθνή σκηνή και είναι σημαντικό να συμμετέχει η Κίνα, οι αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το θέμα είναι επίσης να καταλήξουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα και σε σχέση με τις περιφερειακές δομές και άκουσα εγώ και για το Ευρωπαϊκό ETS και για τα περιφερειακά προγράμματα και σχήματα είναι κάτι το οποίο αποτελεί θα έλεγα την βασική ανησυχία της ΙΚΑΟ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΙΚΑΟ, ξέρετε, είναι ρόλος παρατηρητή και τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν συνεργάζονται μαζί μας ακολουθούμε θα έλεγα μια ενιαία αντίληψη, αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι κοινέ ευρωπαϊκές θέσεις. Εμείς περιμένουμε λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν με ρωτάτε για τα ποσοστά, τα θέματα μέχρι τώρα είναι αρκετά έφραστα Το θέμα είναι ποιες χώρες θα συμμετέχουν και δεν θα ήθελα εγώ να κάνω τώρα προβλέψεις αστήρικτες. Το θέμα είναι να καλύψουμε περιβαλλοντικά τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τώρα, για τις ΙΠΑ και για την αποκλειστικότητα. Εμείς είχαμε κάποιες θετικές συζητήσεις με τις ΕΠΑ τους προηγούμενους μήνες και κατανοούμε τώρα καλύτερα το πού ε, βρισκόμαστε ο καθένας. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτής της αμοιβαία κατανόησης θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και ελπίζω να καταλήξουμε κάπου που θα συμφωνούμε και εμείς για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα στην εφαρμογή των εσωτερικών συστημάτων. Τώρα για τα credits. Εμείς συνειδητοποιούμε τη σημασία του προβλήματος και σε σχέση με την Συμφωνία των Παρισίων και σε σχέση με τα νέα credits. Είναι σαφές σε σχέση με το πρώτο κομμάτι ε, ποια είναι η θέση μας. Σε σχέση τώρα με το ευανάγνωστο των κριτηρίων και των αντισταθμισμάτων, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει την επόμενη Γενική Συνέλευση. Και το είπα πριν αυτό, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Εμείς θέλουμε ε, τα credits τα οποία να είναι πιστοποιημένα από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι βασικά η θέση μας. Σχετικά με μια ισχυρή διαδικασία αναθεώρησης. Αυτή είναι η ερμηνεία την οποία δίνουμε και εμείς στην πρόταση ψηφίσματος. Αλλά όπως είπα έχουμε να κάνουμε με work in progress. Τα πράγματα συνεχίζουν να εξελίσσονται και για μια ακόμη φορά οι λεπτομέρειες για τα μητρώα, τα συστήματα παρακολούθησης, όλα αυτά είναι τμήματα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από την Γενική Συνέλευση μετά την κατάληξή της σχετικά με την ποιότητα των αντισταθμισμάτων, ε, τις περιφερειακές προβλέψεις και την πιλωτική φάση. Κοιτάξτε, ο όρος πιλωτική φάση στην ουσία είναι αυτό που θα λέγαμε μία ρήτρα opt-in, μία ρήτρα εθελοντικής συμμετοχής. Αυτό το οποίο έχει σημασία στην παρούσα φάση είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των κρατών τα οποία καλύπτονται, ανεξαρτήτως του τίτλου του σχήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θέλει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα από το 2021. Όμως θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και με τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουμε αλλάξει μέχρι τώρα τις φιλοδοξίες μας γύρω από το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατόν. Η προσπάθεια συνεχίζεται, πάντως και δεν θέλω να προκαταλάβω την έκβαση. Αλλά <coughs> νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, συνεχίζονται. Σας έδωσα την εικόνα, σας έδωσα το τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρθηκα σε αυτό και στα της Γενικής Συνέλευσης ε, σύντομα. Να θυμίσω επίσης ότι η συνεργασία με τους εταίρους μας είναι κάτι το καθοριστικό. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα με τα opt Στόχος μας θα πρέπει να είναι να προσπαθήσουμε να βεγιστοποιήσουμε την κάλυψη και να συμπεριλάβουμε όλες τις σημαντικές αεροπορικές χώρες. Σημαντικές ενώ στον τομέα, στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας. Έτσι θα αυξήσουμε την κάλυψη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε επίσης και με τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με στρέβλωση του ανταγωνισμού, πάντως θα το παρακολουθήσουμε από κοντά. Θα αναφερθούμε γύρω από αυτό το θέμα και ε, στις ε, άλλες χώρες και στα άλλα μέρη και θα δούμε αν μπορούμε να ε, κάνουμε κάτι περισσότερο. Έχει επίσης σημασία αυτό που είπα προηγουμένως, ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε όλες οι χώρες, οι σημαντικές για την πολιτική αεροπορία, να συμμετέχουν εθελοντικά, θα πρέπει τα μεγάλα διεθνή ε, σημεία ε, επαφής των πτήσεων, τα μεγάλα hub δηλαδή, να καλυφθούν, τα μεγαλύτερα αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι προσπάθησα να καλύψω τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες απαντήσεις. Τέθηκε επίσης και ένα θέμα για το πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ. Εμείς περιμένουμε ένα κείμενο ε, να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑΟ το ταχύτερο δυνατόν. Ακόμα και σήμερα έχουν καθυστερήσει η συνάντηση έγινε την Παρασκευή, εμείς περιμέναμε νωρίτερα να βγούνε, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη βδομάδα θα τελειώσει η ιστορία και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των αποφάσεων και δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες και για παρανοήσεις. Μέσα σε 24 ώρες. Θα ήθελα επίσης να δούμε ποιο είναι το τελικό κείμενο μετά από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Κατανοώ τις θέσεις οι οποίες ε, έχουν εκφραστεί. Κατανοώ την ανάγκη να είναι πολύ φιλόδοξο το μέτρο αυτό, το νέο, το GMBM, οι διαπραγματεύσεις οι διεθνείς αυτές όμως όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερος περίπλοκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες που ελπίζουν όλοι στο να υπάρξει μια ευτυχής κατάληψη. Η επιλογή μας δεν μπορεί να είναι η αποτυχία. Πρέπει να προωθήσουμε τα σφαιρικά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει νομίζω να είμαστε όσο περισσότερο φιλόδοξοι γίνεται. Thank you very much for your... Ευχαριστώ πολύ κύριε Ολολέη. Για τα λεγόμενά σας μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρας διάταξης που είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωμοδότηση του κυρίου Ζάνη για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη από την Επιτροπή Μεταφορών και δίνω μέσω στο λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε σίγουρα όλοι σας, οι δρομοδοτήσεις έχουν ένα αυστηρό περιορισμό σε αριθμό χαρακτήρων. Και γι' αυτό στο σύντομο αυτό σχέδιο γνωμοδότησης προσπάθησα να εστιάσω στα πιο σημαντικά θέματα της, ε, των αερομεταφορών από την οπτική γωνία του περιβάλλοντος. Θέλω λοιπόν να σταθώ στα τωρινά και τα προβλεπόμενα επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος από τον αεροπορικό κλάδο και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό πλαίσιο Επομένω, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησή μου μπορεί να θεωρηθεί μονάχα, θα πρέπει να το θεωρήσετε μονάχα ω ένα αρχικό σημείο εκκίνησης. Είμαι έτοιμο να καλοδεχτώ τα σχόλιά σα και τι τροπολογίε. Θα ήθελα και ο ίδιο να εξελίξω περισσότερο ορισμένα σημεία με τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Αερομεταφορές είναι βέβαια ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει σαφείς επιπτώσεις για το περιβάλλον. Δυστυχώς, εδώ δεν αναφέρεται στην Συμφωνία των Συμβαλωμένων Μερών ή διεθνείς αερομεταφορές, αλλά είναι τεράστια η συμβολή του τομέα αυτού, γιατί χωρίς να, τις αερομεταφορές δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Προβλέπετε ότι οι εκπομπές από τις αερομεταφορές θα είναι 5 φορές, 7 φορές μεγαλύτερη το 2050 από ότι το 1990 παρά το ότι κάθε νέα γενιά αεροσκαφών μειώνει τις εκπομπές κατά 15 με 20%. Ω εκ τούτου χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα για να μην επιδεινώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. την μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, την ρήπανση της ατμόσφαιρας κτλ. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών και ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής και της ρήπανσης είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι στο κέντρο της γνωμοδότησής μας. Θα πρέπει να στείλουμε σαφή μηνύματα στην αρμόδια τη της ουσίας Επιτροπή Τραν, αλλά σε τελική ανάλυση και στην Κομισιόν και τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία, τα εξαποστάσεως κατευθυνόμενα ε, αεροσκάφη, τη χρήση βιοκαυσίμων κτλ. Θέλω να εκφράσω λοιπόν και την ανησυχία μου για το γεγονός ότι βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται δεν έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Γεωργίας να διατυπώσει κάποια γνωμοδότηση. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να κινητοποιηθούν για να υπάρξει και γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας. Χωρίς λοιπόν έρευνα και ανάπτυξη, οι βελτιώσεις στον τομέα των αερομεταφορών δεν θα προκύψουν. Είμαι πεπισμένο ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα αυτό. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την προστασία των καταναλωτών. Υπάρχει μια ανάγκη βέβαια να μειώσουμε το άχθος της ρύθμισης, να βελτιώσουμε την ικανότητα και τις υποδομές και στο έδαφος και στον αέρα, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγάλη έμφαση στην προστασία των καταναλωτών. Θα κλείσω λοιπόν εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη μας συζήτηση για το θέμα αυτό και προσβλέπω στις προτάσεις σας, στις τροπολογίες σας και στη συνεργασία βέβαια με τους σκιώδεις Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκαρντί, Η κυρία Γκαρντίνη, εκ Πατριτσέλο. Ευχαριστώ. Εδώ έχω το σημείωμα που μου έδωσε ο συνάλφος Πατριτσέλο που δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θέλουμε να προχωρήσει η έκθεση αυτή για τους λόγους οι οποίοι ήδη εκφράστηκαν. Ε, η πολιτική αεροπορία αντιπροσωπεύει αγαπητοί συνάδελφοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ισχυρό θα έλεγα μέσο οικονομίας, οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. Ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας παρέχει θέσεις απασχόλησης σε δύο περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ε, κύκλος εργασιών 110 δις κατέτος. Το τελευταία 20 ετία η πλήρης φιλελευθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς όπως και η ανάπτυξη της ζήτησης ε, μας οδήγησαν σε μια ουσιαστική ανάπτυξη των αερομεταφορών με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω προόδου. Θεωρείται ότι το 2035 οι αερομεταφορές στην Ευρώπη θα πρέπει να φτάσει στο, στους 14,4 ε, ε, εκατομμύρια πτήσεις, δηλαδή μια τρομακτική αύξηση σε σχέση με το 12. Γι' αυτό λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας που θα επιτρέψει στον τομέα αυτό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και την αποδοτικότητά του είναι μια καλή πρωτοβουλία και θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή οικονομία, θα ενισχύσει τη βιομηχανική βάση και θα συνεισφέρει στην ηγέτιδα θέση της Ένωσης. Ένας ισχυρός τομέας ο οποίος να καλύπτει και ε, την παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο την Ευρώπη, και με στόχους αηφορίας είναι ένα πλεονέκτημα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες γιατί θα τους παρέχει περισσότερες δυνατότητες συγκοινωνίας με καλύτερες τιμές και με καλύτερη ασφάλεια. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν χαιρετίζω εγώ την πρόταση την οποία προτείνει ο συνάδελφος ε, που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Χάρη και στην συζήτηση που κάνουμε τώρα και στις εφαρμοστικές προτάσεις οι οποίες μαζί με τους συναδέλφους θα κατατεθούν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση λοιπόν και θέση η οποία θα πρέπει να είναι και αρκετά ε, φιλόδοξη. Thank you very much. And now Mr. Eh, Ο κύριος Τόρμαν. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή φυσικά τον κύριο Σάνη για το έργο του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ε, εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα, διεθνή ανταγωνισμό, δικαιώματα επιβατών, τα αερολιμενικά τέλη. Έχω την αίσθηση μερικέ φορές ότι τα προβλήματά μας συσσωρεύονται. Επίσης το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ειδικευμένο προσωπικό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη μια γενική και ευρεία στρατηγική. Εδώ τώρα εξετάζουμε το περιβαλλοντικό σκέλος αυτής της στρατηγικής. Ο εισηγητής μας ε, ε, μας λέει ότι ο αεροπορικός κλάδος ε, εξαιρείται από τις συμφωνίες των Παρισίων, αλλά και άλλοι κλάδοι πλήττονται από τις απαιτήσει που έχουμε σε περιβαλλοντικά θέματα και θεωρώ ότι όλοι οι τομεί και η αεροπορία θα πρέπει να συμβάλλουν στην αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών γιατί και η αεροπορία συμβάλλει ε. στις κλιματικές αλλαγές. Βέβαια, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πια όλο και πιο φθηνά. Θα πρέπει λοιπόν να, σκεφτούμε πώς θα συμβάλλει και η αεροπορία περαιτέρω. Πάντως ξεκινήστε με καλές βάσεις. Ευχαριστώ κύριος Έκχαουτ. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι λακωνικός ε, γιατί μακρηγόρησα στο προηγούμενο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί δεδομένου του περιορισμού στην έκταση της ε, γνωμοδότησής του τουλάχιστον επισήμανε τα βασικά ζητήματα. Και με τις τροπολογίες μας εμείς απλώς θα συμπληρώσουμε κάποια θέματα, κάποιε λεπτομέρειες σε ζητήματα που ήδη είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, γιατί είναι σημαντικό από περιβαλλοντική άποψη. Θα καταθέσουμε και τροπολογίε όχι μόνο για το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί όταν μιλούμε για την αεροπορία δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο, με το, μόνο στο διοξίδιο του άνθρακα, παρόλο που το τονίζουμε συχνά. Επίση, είπατε ότι θα συνεχίσουμε το δικό μα ε, σύστημα εμπορία εκπομπών ε, όσο δεν έχουμε παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Ε, ίσως πρέπει να αναδιτυπώσουμε το σημείο αυτό μετά και την προηγούμενη συζήτηση, γιατί το μόνο κριτήριο δεν είναι να έχουμε παγκόσμιο απλώς αγοροκεντρικό μέτρο. Θέλουμε ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο μέτρο. Αλλιώς να συνεχίσουμε το δικό μας σύστημα εμπορίας εκπομπών όσο δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό ή αποδοτικό αγοροκεντρικό μέτρο που αυτή τη στιγμή εξετάζεται στον ΙΚΑΟ. Αυτά και θα υποστηρίξουμε την γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρος κ. Φάντερ. Κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο μας προτείνεται, το έγγραφο που μας προτείνει η Κομισιόν, μου φαίνεται ότι είναι μια ισχυρή βάση η οποία θα επιτρέψει τη μείωση του, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις αερομεταφορές. Αλλά τίθεται και το θέμα της ανταγωνιστικότητας αυτού του τομέα. Είναι σημαντικό θέμα γιατί απασχολεί εκατομμύρια ο τομέας των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Είναι σημαντικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την προβληματική του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα <clears throat> στην υποστήριξη που θα πρέπει να δώσουμε στην εφαρμογή των ενιαίων εθέρων στην Ευρώπη και στα ερευνητικά σχέδια όπως το ΣΕΖΑΡ για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Γιατί μόνο με το να βελτιστοποιήσει τα σχέδια πτήσης και την μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα ελαφραίνοντας παράλληλα το βάρος προς το περιβάλλον. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν την εφαρμογή του προγράμματος ΣΕΖΑΡ. Κλείνω λέγουσα ότι η υποστήριξη στην έρευνα στον αεροναυπηγικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να δράσουμε στην πηγή των ε, αερίων του θερμοκηπίου και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο αεροναυπηγικός τομέας για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ε, απόδοση των κινητήρων των αεροσκαφών. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο Πρόεδρος. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε και την Κομισιόν, την, την κυρία Πόρτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι και όλη την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χαίρεται που βλέπει την Επιτροπή Περιβάλλοντος να εκφράσει την απόψή της για ένα τόσο σημαντικό θέμα για την πτυχή του περιβάλλοντος ε, στη στρατηγική για τις αερομεταφορές που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρόμαστε επίσης που ακούμε ότι τα μέλη της Επιτροπής σας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των αερομεταφορών στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ήταν και το πρώτο στοιχείο της ανακοίνωσης της Κομισιόν και εξακολουθεί να είναι από τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλουμε να υπογραμμίσουμε σήμερα. Προσβλέπουμε να δούμε <clears throat> πώς θα τροποποιηθεί περαιτέρω το κείμενο αυτό από την ε, Επιτροπή σας για να αρρωγήσει την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ακούσω τώρα και τον εισηγητή, εάν θέλει να λάβει για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο εισηγητή. Πιστεύω ότι ε, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ μας, δεν είναι αφιλεγόμενο το θέμα και χαιρετίζω την προσήλωση όλων των συναδέλφων και ιδιαίτερα των σχεδόν εισηγητών που φάνηκε από τη συζήτηση. Περιμένω με χαρά τα σχόλια και τις τροπολογίες τους και προσβλέπω στην εκπόνηση μιας αξιόλογης γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα μόνο. Προθεσμία για τις τροπολογίες 6 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 29 Σεπτεμβρίου. Στην Επιτροπή Μεταφορών η ψηφοφορία θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου για να πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Και περάμε τώρα στο επόμενο θέμα. πρόκειται για την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία των Παρισίων που εγκρίθηκε στα πλαίσια τη Σύμβαση Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Θα γίνει συζήτηση του σημείου αυτού από κοινού με το σημείο 9 την διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το COP22 του 2016 στο Μαρακές και να δώσω πρώτα το λόγο στον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι ο εισηγητής για το 8 και θα τα, σας τα πω στα Ιταλικά. Η συμφωνία λοιπόν των χωρών αυτών είναι μια θα έλεγα πολύ σημαντικό βήμα στα πλαίσια της καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Η πρόταση είναι φιλόδοξη, ισορροπημένη και νομικά δεσμευτική. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε κομβικό ρόλο για την επίτευξη της συγκεκριμένης συμφωνίας. Νομίζω ότι είναι ε, γνωστή σε όλους οι όροι της συμφωνίας αυτής. Τους επαναλαμβάνω πάντως, μακροπρόθεσμη μορφή προγραμματισμού, να φτάσουμε ε, σε επίπεδα τα οποία να μην ξεπερνούν τους δύο βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ενίσχυση ε, της, ε, των μέτρων τα οποία φιλοδοξούμε να πάρουμε έτσι ώστε να έχουμε σύντομα ένα συνολικό απολογισμό γύρω από τις εκπομπές και κυρίως μια ιδιαίτερη συμμετοχή των χωρών κάτι το οποίο αποτελεί μια καινοτομία σε σχέση με τις προηγούμενες συμφωνίες. Η Συμφωνία των Παρισίων καλύπτει όλες τις μεγάλες χώρες, και όχι μόνο τμήμα Σήμερα ασχολούμεθα με την πρόταση επικύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα υπεγράφει η συμφωνία από πλευρά Συμβουλίου και Επιτροπής στις 22 Απριλίου στη Νέα Υόρκη. Θα τεθεί σε εφαρμογή την 30η μέρα μετά από το 55% των συμμετεχόντων και από το 55% μάλλον της 100% των αυτών που εκπέμπουν τέτοιου είδους αέρια θα πρέπει να έχουν επικυρώσει. 188 χώρες έχουν υπογράψει και 26 έχουν καταθέσει τα μέσα και τις διαδικασίες επικύρωσης. Η διαδικασία εξελίσσεται με αργή ταχύτητα. Στο εσωτερικό της Ένωσης τρεις χώρες έχουν ολοκληρώσει την επικύρωση, Ουγγαρία, Αυστρία και Γαλλία. Δεν έχουν όμως καταθέσει το αποτέλεσμα της επικύρωσης αναμένοντας και τις υπόλοιπες χώρες και το σύνολο της Ένωσης. Μέχρι τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει τα μέσα επικύρωσης δεν καλύπτουν παρά μόνο το 1% των σφαιρικών εκπομπών. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή για μικρές χώρες, από αυτές οι πιο μεγάλες είναι το Καμερούν, η Βόρεια Κορέα, το Περού και η Νορβηγία. Ε, ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε λειτουργία το 2016 ε, και θέλουμε να παλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία χωρίς την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θα αμφισβητήσει την ηγετική θέση της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να καλέσουμε το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι διαδικασίες επικύρωσης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο να γίνουν πριν το, 16, πριν το τέλος του 2016. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή των υποχρεώσεων μας σε εθνικό επίπεδο από το 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ένα φιλόδοξο θα έλεγα πρόγραμμα έτσι ώστε να καλύψουμε τουλάχιστον το 40% μέχρι το 2017. Η διαδικασία επικύρωσης λοιπόν θα στείλει θα έλεγα ένα ισχυρό μήνυμα, θα αποδείξει την ηγετική θέση της Ένωσης και θα αποδείξει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Είναι μια βασική προτεραιότητα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να στηρίξετε λοιπόν παρακαλώ την πρότασή μου στο Συμβούλιο να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων και να τονίσουμε τις διαδικασίες εθνικής επικύρωσης, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επικύρωσης και να καταθέσουμε στα Ηνωμένα Έθνη τα απαιτούμενα μέσα, τα νομικά, πριν από το τέλος του έτους. Τώρα θα ξεκινήσει η κοινή συζήτηση και θα δώσω το λόγο και στους συναδέλφους οι οποίοι υποστηρίζουν την πρόταση ψηφίσματος και για την COP22 στο Μαρακές. Παγνιό. Κύριε Πρόεδρε, και συνάδελφοι, όπως μας είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, εννέα μήνες μετά την COP21 στο Παρίσι, ήρθε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να περάσουν από τα λόγια στα έργα. Και ως συγητής ε, του ψηφίσματός μας για την COP21, διαπιστώνω ότι οι ολιγορίες ε, στη διαδικασία κύρωσης σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ ενισχυτικές. Εγώ τουλάχιστον ανησυχώ τα μάλα, γιατί κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ξεκινήσει νομοθετικές διαδικασίες που μάλιστα έχουν ακολουθήσει την αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή που ακολουθούσαν οι υποσχέσεις των ίδιων κυβερνήσεων. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και χώρες που δεν είναι ακόμη σε θέση να μας κοινοποιήσουν το χρονοδιάγραμμά τους ε, για να ε, περιορίσουν τους κλάδους ε, του άνθρακα που συμβάλλουν στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα το, διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει τουλάχιστον 55 χώρες ε, να το κυρώσουν με πάνω από 55% του συνόλου των ε, παγκοσμίων εκπομπών, αλλά ακόμη πόρα απέχουμε από αυτό το στόχο, γιατί οι 26 χώρες που αναφέρθηκαν, που ξεκίνησαν τη διαδικασία κύρωσης, ε, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε υπάρχει πια επιτακτική ανάγκη και μάλιστα πριν την COP22 του Μαρακές, πριν τις 7 Νοεμβρίου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούμε όπως το κάναμε και για το Παρίσι και να περάσουμε, επαναλαμβάνω, από τα λόγια στα έργα. Γιατί ε, είναι, αν μη περίεργο, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιοχές που περισσότερο συμβάλλουν στην αύξηση του διοξίδιου του άνθρακα, να μην έχουν κυρώσει ακόμη αυτή τη συμφωνία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κυρώσει, μπορεί από μόνη της να κυρώσει τη Συμφωνία των Παρισίων, ε, ως νομική οντότητα και να μην περιμένει από τις μεμονωμένες χώρες μέλη να το κάνουν. Και χθες ε, μίλησα με τη Σεγκολέν Ρογιάλ ε, στο τηλέφωνο και μου είπε ότι από νομική άποψη δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιμένει την απόφαση κύρωση των χωρών μελών, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της να προβεί στην κύρωση. Και όπως μας είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος, δηλαδή, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε εμείς και τα κοινοτικά μας θεσμικά όργανα και να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και μάλιστα θα καταρτήσουμε αυτό το ψήφισμα που θα εγκριθεί στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου και με το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να διατρανώσουμε την άποψή μας και να γίνει αυτή η πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου ορόσημο και σημείο αναφοράς για το Συμβούλιο, ώστε και αυτό να επισπεύσει τις διαδικασίες και να λάβει αποφάσεις σε συνεργασία με εμάς και το την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπει επιτέλους αυτή η υπογραφή της κύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων και ζήτησε από τον πρόεδρο Σούλτς να αξιοποιήσει αυτή την ολομέλεια για να καλέσει την Σεγκολέ Ροαγιάλ που ήταν πρόεδρος της COP21 στο Στρασβούργο για να εκφωνήσει ομιλία. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το δεύτερο ψήφισμα που αφορά την προετοιμασία για την COP22 στο Μαρόκο. Έχω συνυπογράψει πολλές τροπολογίες με τον Γιώ Λάινεν που δυστυχώς απουσιάζει σήμερα και τη Σιμώνα Μποναφέ ζητώντας ε, κάποια κρίσιμα σημεία να τα αναφέρουμε και στο ψήφισμα. Για παράδειγμα, τη δημιουργία καινοτόμων μέσων χρηματοδότηση για να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, όπω την θέσπιση ενό φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τον προσδιορισμό μια ε, οριακή τιμή ε, για τον τόνο ε, του διοξιδίου του άνθρακα, ποσόστοση άνθρακα, επίση θέσπιση πραγματικής κυκλικής οικονομίας και ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί αυτή είναι η πρόκληση που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Επίσης, ε, κατάργηση των επιδόσεων στον τομέα ορυκτών ε, ε, καυσίμων για να εγκαταλείψουμε σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών και της γεωργίας, στόχοι 2020-2030. Επίσης, 100 δισεκατομμύρια το χρόνο υποσχέθηκαν οι αναπτυγμένε χώρες μέσω του Πράσινου Ταμείου να χορηγήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ακολουθήσουν αυτούς τους στόχους. Επίσης, ε, ε, η Αφρική έχει ένα τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δυστυχώς ε, παραμένει αναξιοποιητό. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Επίσης, ε, να αναγνωρίσουμε διεθνώς το καθεστώς του περιβαλλοντικού πρόσφυγα, αναγνωρίζοντας τις συνέπειες που έχει μόλις του περιβάλλοντος στις μεταναστευτικές ουρές. Αυτά θα προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα για την COP22, γιατί νομίζω ότι επήγει το θέμα και θα πρέπει επιτέλους να θεσπίσουμε κοινοτική νομοθεσία σχετικά και μάλιστα σχετικά γρήγορα και στα τέλη του έτους και καθ' την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο Τζοβάνι Λαβία για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων και θέλω να ευχαριστήσω και τις άλλες πολιτικές ομάδες που υποστήριξαν την έκθεση της Επιτροπής μας, γιατί με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα για την κύρωση της συμφωνίας αυτής. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει. Για το ψήφισμα τώρα για το Μαρακές, εγώ είμαι αρμόδιος από την πλευρά του ΕΛΚ, πιστεύω ότι αυτή η αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή να υπάρξει συνένεση μεταξύ κομμάτων αλλά και μεταξύ επιτροπών. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπήρξε μια έκθεση από την Επιτροπή Βιομηχανίας από όλα τα κόμματα και αυτό πράγματι αν το υποστηρίξουμε θα βελτιώσει την δυνατότητα ε, ουσιαστικής συνένεσης στην Ολομέλεια. Αν υποστηρίξουμε όλη την πρόταση της Ήταν μια μεγάλη επιτυχία η συνδιάσκεψη των ε, Παρισιών ήταν ένα μεγαλούργημα σε διπλωματικό επίπεδο, χάρη και στη Γαλλική Προεδρία κυρίως, αλλά και πολλούς άλλους. Θα πρέπει να είναι σαφέ όμως ότι όλες οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν στο Παρίσι δεν είναι επαρκείς για να επιτευχθεί ο στόχος της μη αύξησης πέραν των δύο βαθμών Κελσίου της θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Πώς θα πετύχουμε λοιπόν αυτό το στόχο. Είναι δύσκολο βέβαια πια να μιλάμε για μόνο αύξηση 1,5. Αυτό είναι ευχή έργο. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε καν το στόχο 2 βαθμών, δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπονομεύσουμε την προσπάθειά μας. Αλλά είναι σαφές ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να γίνει από όλους, δεν μπορεί να την κάνει μόνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να ξεπεράσει τους στόχου που έχουν τεθεί. Αυτό όμω θα είναι κενό νοήματος αν δεν υπάρξει συνολική συμφωνία με όλους τους άλλους διεθνείς εταίρους της. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μετά από τις εκλογές στις οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αν κερδίσει ο Τραμπ τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αν κερδίσει όμω η Κλίντον θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Επίση πρέπει να δούμε και με την Κίνα πώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γι' αυτό θέλω να υποστηρίξω όλε αυτέ τι τροπολογίε οι οποίε υποστηρίζουν ένα διεθνέ γίγνεσθε. Είναι δύσκολο να υπάρξει κατά την άποψή μας μια περαιτέρω βελτίωση των στόχων από την Ευρώπη και μόνο θα πρέπει να συμπορευτούμε με τη διεθνή κοινότητα. Για μας, για το ΕΛΚ, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμποδίσουμε και την λεγόμενη διαρροή άνθρακος, δηλαδή την ε, μετακίνηση επιχειρήσεων για να αποφύγουν τους στόχους αυτούς. Θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία για όλα αυτά τα θέματα, επομένως και ένα σωστό μείγμα ευφυών εργαλείων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κλιματικοί πρόσφυγες τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει μια καλή συμβαστική λύση στο κείμενο που έχουμε εγκρίνει πέρσι και πρόπερσι είναι επίσης ευκταίο να υπάρξει και ένα νομικό καθεστώς για τους κλιματικούς πρόσφυγες. Αυτό στην τρέχουσα χρονική στιγμή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρουμε ποιες συνέπειες θα προκαλούσε. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στο κείμενο που έχουμε τώρα ως βάση ή αλλιώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία 170 της Judy Girling, η οποία τονίζει καλύτερα τα θέματα αυτά, αλλά το να ζητήσουμε μια νομική ρύθμιση του καθεστώτος των κλιματικών προσφύγων, αυτό θα μας οδηγήσει σε μεγάλες δυσκολίες στην Ολομέλεια. Η διαδικασία τώρα για την εκπόνηση αυτού του ψηφίσματος ε, δεν είναι η καλύτερη γιατί έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου θα προτιμούσα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και για τις χωριστές ψηφοφορίες και τις ε, ψηφοφορίες κατά τμήματα εκπνέει προθεσμία αύριο το πρωί ή μάλλον απόψε το βράδυ από ό,τι κατάλαβα. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να την καθυστερήσουμε λιγάκι αυτή την προθεσμία Όλοι γυρίσουμε από τις διακοπές και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πάρα πολύ σφιχτές προθεσμίες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο της Επιτροπής και τη Γραμματεία να δουν αν μπορούμε <clears throat> να κάνουμε μια ε, αναβολή αυτής της προθεσμίας μέχρι τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για τις ε, χωριστές ψηφοφορίες και τις ε, ψηφοφορίες κατά τμήματα. Θα επιτρέψει στις ομάδες να έχουν μια καλύτερη διατύπωση της θέσεως. Αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν για το διαδικαστικό θέμα, για τη διαδικαστικό επίπεδο. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η ομάδα του ΕΛΤ θέλει να αποτρέψει την λεγόμενη διαρροή άνθρακος, αλλά παρόλα αυτά υποστηρίζει μια φιλόδοξη πολιτική στα κλιματικά θέματα, μαζί με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Βιομηχανίας, ιδίως τον Ιβο Μπέλετ, έχουμε εργαστεί από κοινού και θέλουμε να υπάρξουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της μόνωσης των κτίριων. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσα από την ε, εφαρμογή της οδηγίας που προτείνει η Κομισιόν για την ενεργειακή απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τον ζητήσει πάντα να υπάρξει ένα στόχος 40%. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο βρίσκονται μονάχα στο 27% για την ενεργειακή απόδοση και βρισκόμαστε στο δίλημα ότι με τη σύγκρουση αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι είναι μη ρεαλιστική η, ο στόχο, ρεαλιστικός στόχος 40%. Γι' αυτό έχουμε την τροπολογία 220, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει μια συμβαστική λύση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων <clears throat> θεσμικών οργάνων. Μπορούν δηλαδή και οι δύο πλευρές να βρουν κάποια ενδιάμεση λύση. Σας παρακαλώ λοιπόν να δείτε την τροπολογία 220 και αν μπορείτε να την υποστηρίξετε, γιατί με μια αύξηση της ενεργειακής ε, απόδοσης θα προωθήσουμε μια φιλόδοξη πολιτική για, τα κλιματική, για την κλιματική αλλαγή, αλλά και συγχρόνως θα αποτρέψουμε την μετακίνηση επιχειρήσεων, τη λεγόμενη διαρροή άνθρακος και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε και την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ευρωπαϊκή μας ε, ε, ήπειρο χωρίς να υπάρξει μετακίνηση επιχειρήσεων και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση. Τα 27% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι πολύ λίγο. Το 40% για τα άλλα θεσμικά όργανα και για το ΕΛΚ είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Έχω καταθέσει αυτή την τροπολογία να μείνουμε στο 30% με τη δυνατότητα να φτάσουμε στο 40% και θα χαρώ πολύ αν υποστηρίξουν την τροπολογία μου αυτή και οι άλλοι συνάδελφοι. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Νομίζω ότι όλοι περίπου συμφωνούμε και για τις διαδικασίες επικύρωσης. Η δική μου εμπειρία λέγει ότι ίσως τα πράγματα να είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι περιγράφονται τώρα. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές είναι πιο φιλόδοξη από τη συμφωνία, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, προβλήματα, εκτός και αν υπάρχουν ευρύτεροι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα. Το θέμα λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία επικύρωσης και δεν ξέρω αν νομικά στέκει το να επικυρώσει η Ένωση χωρίς να έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη-μέλη ή ακόμα και αν στέκει νομικά πολιτικά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Συνεπώς λοιπόν εμείς σαν βουλευτές πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες τις οποίες έχουμε Είναι μια συμφωνία ιστορική στην οποία έχουμε καταλήξει υπό την καθοδήγηση μιας μεγάλης ε, ευρωπαϊκής χώρας. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία όμως. Και είναι κατανοητό ε, το ότι κάποια κράτη-μέλη δεν ε, επιθυμούν στη συγκεκριμένη περίπτωση μια σφαιρική απόφαση να καλύψει τις δικές τους δυνατότητες και αρμοδιότητες. Εν πάση περιπτώσει, ας μην ε, μεγαλοποιούμε το θέμα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πλήρως υπέρ της συμφωνίας αυτής και θα πρέπει αυτό και μόνο να μας ε, οδηγήσει σε μια λύση. Για τη δεύτερη έκθεση τώρα, Οι διαπραγματεύσεις ε, καθυστέρησαν γιατί μεσολάβησε ο χειμώνας, μετά ήρθαν οι καλοκαιρινές διακοπές, Πάντα υπάρχουν τέτοιου είδους εξηγήσει. Πάντως θέλουμε να συνεργαστούμε γρήγορα έτσι ώστε να καταλήξουμε στις συμβιβαστικές προτάσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με αυτό. Ξέρω ότι πολύ συχνά υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να δω εδώ είναι να είναι ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη πρόταση, ένα ξεκάθαρο ψήφισμα, να μην το φορτώσουμε με διάφορα καλούδια δεξιά και αριστερά. Ε, έτσι θα ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας για το Μαρόκο, αλλά δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου όλοι θα βάζουν τις δικές τους επιθυμίες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γερμπάντη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της διαχείρισης της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Γιατί αυτό με προβληματίζει αρκετά. Φυσικά έχουμε ένα πολύ θετικό σενάριο με μια ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας χάρη σε μεγαλύτερη συγκέντρωση μα στο στόχο της ε, οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο και κάπως πιο απότομα. Και προς το παρόν θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η διαχείριση που κάνουμε και πολύ φοβάμαι ότι θα ισχύσει το αρνητικό σενάριο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε φέτος το Φεβρουάριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και ε, μάλιστα έγινε δύο μήνες μετά το Παρίσι η δημοσίευση και γι' αυτό δεν ε, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και περιγράφει αυτά τα δύο σενάρια και τους κινδύνους ε, να υλοποιηθεί το αρνητικό ε, και απότομο σενάριο Επίσης, ε, έχουμε και το θέμα των συστημικών κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ε, ξαφνική ε, αναβάθμιση στοιχείων ενεργειοβόρων με υψηλά ποσοστά άνθρακα. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τους ενδεχόμενους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με μια απότομη μετάβαση και επίση τι μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε για να αποσοβήσουμε αυτού του κινδύνου. μια στρατηγική για τα μέσα του αιώνα με μηδενικές εκπομπές και να βρούμε ένα ε, πιο αποτελεσματικό δρόμο προς ε, μια τέτοια οικονομία. Φαίνεται πολύ τεχνικό, ακούγεται πολύ τεχνικό και αρκετά απόμακρο, αλλά εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις, αλλά όλο και αναβάλουμε προς το μέλλον τα πιο σημαντικά θέματα. Και οι εμπειρογράμμονες θεωρούν ότι θα είναι τεράστιοι κίνδυνοι και μεγάλες ε, οι οικονομικές ζημίες ε, και μάλιστα δυσβάσταχτες. Θα ήθελα λοιπόν να επιζήσω την προσοχή σας ε, σε αυτά τα δύο στοιχεία, θα τα καταθέσω και στις τροπολογίες μου και ελπίζω να τα σχολιάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ικ Άουτ. Σας ευχαριστώ και εγώ πρώτα απ' όλα για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Είναι λίγο πιο σημαντικό αυτό από ότι το έθεσε η Τζούρι Γκέρλινγκ. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο και πολιτικό θέμα για την Ευρώπη. Όταν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ο παγκόσμιο ηγέτης για την κλιματική αλλαγή και εάν μετά από μια τέτοια δήλωση δεν είμαστε οι πρώτε χώρε που θα κυρώσουν αυτή τη συμφωνία και θα την εφαρμόσουμε, θα είναι ένα έσχο για την Ευρώπη. Χαίρομαι που η Κομισιόν υπέβαλε πολύ γρήγορα μια πρόταση μετά από την επίσκεψη του κ. Γιούγκερ στην ε, Ιαπωνία και η G8 και G7 του είπαν, ξέρετε, η Ευρώπη ίσως μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα. Χαίρομαι λοιπόν που το έκανε αυτό η Κομισιόν και ελπίζω ότι και το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει με μεγάλη ταχύτητα το απαραίτητο. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τον κύριο Λαβία στο να αναλάβει αυτή την έκθεση, επειδή έτσι θα πάνε γρήγορα τα πράγματα. Δεν είναι όλες σας οι εκθέσεις τόσο γρήγορες, αλλά αυτή θα είναι. Το πρόβλημα βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε το Ηνωμένο Βασίλειο είπε θα το κάνουμε ASAP, το ταχύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια ευγενική έννοια που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ. Όλοι μας θέλουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι το ταχύτερο δυνατό, αλλά μερικές φορές καθυστερεί αυτό λιγάκι. Προ την Κομισιόν, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι την επόμενη εβδομάδα η Κίνα και οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν την κύρωση για το 2016 και η Βασίλεια το έχει κάνει ήδη, εμείς κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα προς την κατεύθυνση των 55 χωρών που εκπροσωπούν το 55% των εκπομπών. Ποιε είναι λοιπόν οι προοπτικέ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφέτο θα κυρώσουν αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να ξέρω πώ προβλέπετε να γίνει αυτό στα κράτη-μέλη και αν υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε θέλουν λίγο περαιτέρω σπρόξιμο. Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί ξέρουμε ότι κάποιε χώρε πάνε πιο γρήγορα από τι άλλε και ξέρουμε ότι όταν υπάρχει πολιτική θέληση μπορούν να προχωρήσουν κάποιες χώρες με την εξαίρεση του Βελγίου που πρέπει να υπάρξει κύρωση από τοπικά και περιφερειακά κοινοβούλια, αλλά και εκεί μπορεί να γίνει. Και επανέρχομαι τώρα στο ψήφισμα μας για το Μαρακές. Το σημαντικό εκεί είναι να κάνουμε σαφές ότι η διάσκεψη του Μαρακές θα πρέπει να είναι και η διάσκεψη για τη δράση μέχρι το 2020. Έχουμε χάσει από τα μάτια μας την ιδέα ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μέχρι το 2020 και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι στεναρότερη. Η Κομισιόν μιλάει πάντα για την νομοθεσία που υπάρχει για τη δράση μέχρι το 2020. Κάπου αναφέρθηκε η Κομισιόν και στο σχέδιο του ΙΚΑΟ στη στοιχείο της δράσης μέχρι το 2020 Ελπίζω ότι τώρα η Κομισιόν έχει τροποποιήσει αυτή τη δήλωση, αλλά οι δράσεις μας μέχρι το 2020 εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές. Και αν δούμε τι άλλο πρέπει να συμβεί, ας είμαστε ειλικρινείς. Ξέρουμε ότι τα σχέδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι προτάσεις συνεισφοράς που πρέπει να γίνουν σαφείς και δεσμεύσεις δεν είναι ακόμα επαρκώς καθορισμένες. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να καταλήξει σε προτάσεις συνεισφοράς που να ξεπερνούν τις μέχρι στιγμής προθέσεις. Θέλουμε οι εθνικές συνεισφορές να ξεπεράσουν τις τωρινές προθέσεις ε, συνεισφοράς. Αν δεν το κάνει λοιπόν αυτό πρώτη η Ευρώπη, πώς θα το κάνουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να το τονίσω και η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανακοίνωση για το χαμηλό ανθρακικό μέλλον μας. Είναι πεπαλαιωμένο, ξεπερασμένο από τα πράγματα. Αυτός ο οδικός χάρτης μιλάει για μείον 8% του 2000, 2050. Μα αυτό είναι το πιο χαμηλό επίπεδο στόχων. Συζητάμε πέραν αυτού στο Παρίσι. Θα πρέπει η Κομισιόν να έρθει με ένα νέο οδικό χάρτη για την μείωση των εκπομπών άνθρακα και ελπίζω να το κάνει τρέχουσα Κομισιόν και όχι η επόμενη Κομισιόν γιατί αυτό θα δώσει και πάλι την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ωραία και μεγαλόσχημα λόγια στο Παρίσι και μετά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και τέλος για την τροπολογία 122 του Πέτερ Λίζε. Συγγνώμη Πέτερ, έχεις χάσει αυτή αυτόν τον αγώνα ήδη πολλές φορές στο παρελθόν. Η πλειοψηφία μας υποστηρίζει τον ενεργειακό στόχο του 40%. Προσπαθήσατε να το αλλάξετε στην Επιτροπή Ήτρε, δεν τα κατάφερες. Και προσπαθήσατε να το κάνεις εδώ. Χαίρομαι για τη συνεπειά σου, αλλά δεν είναι λογικό να ζητάς από την Επιτροπή μας να δεχτεί τις τροπολογίες σου και να υποχωρήσει από αυτό που ήταν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα και πριν από το καλοκαίρι σε μια έκθεση Ήτρε. Υποστηρίζουμε λοιπόν το στόχο 40% για την ενεργειακή απόδοση. Κατανοώ τις προσπάθειες του Πέτερ να βρει κάποιο ενδιάμεσο δρόμο μεταξύ του ΕΛΚ και των υπολείπων, αλλά μέχρι τώρα η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου συγκροτείται χωρίς το ΕΛ και αυτό μερικές φορές είναι και πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αφρόντε θέλει το λόγο. Για την κύρωση. Και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση που έκανε ο πρόεδρος μας. Είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η κύρωση και μάλιστα πριν την επόμενη κόπ. Δεν συμφωνώ ότι δεν επήγει το θέμα. Όχι, σίγουρα επήγει. Δεν ξέρω από τυπική άποψη θα πρέπει τα κράτη-μέλη να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πρώτη την κύρωση ή αν μπορεί αυτόνομα η Ευρωπαϊκή αυτό Ένωση να κάνει την κύρωση. Πάντω, ε, το θέμα είναι κατεπήγον. Θα πρέπει να κυρωθεί και να δώσουμε το μήνυμα ε, και να περάσουμε στι πράξει το συντομότερο δυνατό. Επίση, στο παρελθόν, του προηγούμενου μήνε είδαμε νέες ε, ε, επιστημονικές μελέτες που προτείνουν διαφορετικά μοντέλα, ε, όπως αυτά, όχι μόνο όπως αυτά του πλαισίου του Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχουμε και κάποια οριζόντια μοντέλα που είναι πολύ ενισχυτικά. Και για την ταχύτητα με την οποία δεν αλλάζουν τα πράγματα και για το ποιόν των αλλαγών αυτών. Θα πρέπει εμείς να επιτρέψουμε σε επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε λάβει, αλλά οι διαδικασίες που έχουν ακολουθεί μέχρι τώρα είναι πολύ ανησυχητικές. Για την ίδια την έκθεση, Είδαμε ότι έχουν κατατεθεί σχεδόν 200 ε, τροπολογίες. Αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον προς την θεματολογία τη συγκεκριμένη. Ανακατεύονται πολλά και ετερόκλητα πράγματα εδώ από διαφορετικές πλευρές. Δεν έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά αν θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα ψηφίζουμε υποτίθεται. Σχετικά λοιπόν με την ίδια την έκθεση επαναλαμβάνει ο μιλητής, εμείς θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Το mainstream, έτσι όπως προτείνεται, είναι κάτι το οποίο για μας είναι καθοριστικό. Το θέμα είναι να υπάρχει ε, πίστη στον μηχανισμό ETS, γιατί αλλιώς οδηγούμεθα στην εγκατάληψή του και όχι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να διευρύνουμε δηλαδή το ETS και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλες αγορές. <clears throat> Πέρα από την οικονομική κρίση έχουμε να κάνουμε επίσης και με τις ανανεώσιμες πηγές και στην ενσωμάτωση της διαδικασίας αυτής και στην αγορά ενέργειας. Ο μηχανισμός ETS πάντως, η χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, Έχουμε ε, βιομηχανικούς τομείς οι οποίοι ε, ξεπερνούν τις εκπομπές. Ε, κανονικά οι συνέπειες αυτών των εκπομπών και το κόστος που προκαλούν θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να καλύψουν το κόστος της αρνητικής τους παρέμβασης στο περιβάλλον. Αλλά είναι πολύ διαστραμμένη σε εισαγωγικά αυτή η αντίληψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την μόλυνση από πλευρά των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και να σταθούμε πάντα στις, στα ποσοστά τα οποία έχουμε υποχρεωθεί από μόνοι μας να υιοθετήσουμε. Το θέμα δεν είναι λοιπόν εμείς να επιμείνουμε προς την κατεύθυνση αυτή επαναλαμβάνω το ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στις εκπομπές ε, που προέρχονται από την ε, εντατική κτηνοτροφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάντα σε επικαιρότητα. Ε, Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί να υπάρξει μια σωστή ενημέρωση, μια εκστρατεία ενημερωτική, ε, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει αυτό μέχρι τώρα και αλλιώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους τους οποίους μόνοι μας επαναλαμβάνω έχουμε θέσει. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή σας σε μία από τις πιο παράδοξες πτυχές της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή κάποιες, ε, κάποιοι βιομηχανικοί τομείς που έχουν μεγάλες εκπομπές αλλιώς του θερμοκηπίου έτυχαν μεγάλες προσοχής, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που παράγουν πολλές εκπομπές, οι οποίες κάπου έχουν χαθεί από τον οριζόντα. Σκέφτομαι κυρίως την γεωργία και γενικά την χρήση της γης. Πώς ε, καλλιεργούμε τη γη, πώς προσέχουμε τις, γη, πώς εξετάζουμε τις εκπομπές από τις γεωργικές διαδικασίες. Και αν κοιτάξουμε καλύτερα την χρήση της γεωργικής γης, μπορούμε να προσχωρήσουμε περισσότερο στην αντιμετώπιση των εκπομπών. Ίσως είναι ένας τομέας ο οποίος δεν είναι τόσο ελκυστικός, αλλά η ποιότητα των εδαφών, αν έχουμε πραγματικά μεγάλο οργανικό περιεχόμενο στα εδάφη, τα γεωργικά, τη γεωργική γη, θα μπορούμε να συγκρατούμε περισσότερο άνθρακα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν καλύτερα. Οι συζητήσει λοιπόν που γίνονται για τη γεωργία και την χρήση γης δεν έχουν την ίδια προτεραιότητα όπως ε, οι άλλοι τομείς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη συζήτηση αυτή. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και αυτό είναι από τα καλά της διάσκεψης του Παρισιού ότι η δασοκομεία έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι μονάχα ένα κομμάτι της χρήσης γης. Στην Ευρώπη 10 με 20% των εκπομπών μας ουσιαστικά αντισταθμίζονται από την κατακράτηση άνθρακος από τα δάση μας. Αν μπορούμε λοιπόν να είμαστε πιο ε, αποδοτικοί στην ε, κατασκευαστική βιομηχανία, μπορούμε να μειώσουμε την χρήση άνθρακα. Αν θέλουμε λοιπόν να μετατοπίσουμε την κατασκευαστική δραστηριότητα προς την χρήση ξύλου και όχι μονάχα σιμέντου και χάλιβα που οδηγούν σε μεγάλες εκπομπές ε, του άνθρακος και να κατακρατήσουμε το διοξείδιο του άνθρακος με την ξυλία, αυτό θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην χρήση της γης και τη δασοκομεία <clears throat> δεν είναι αργά για να μπορέσουμε να τονίσουμε τον ρόλο αυτών των δραστηριοτήτων γιατί μπορούν να βοηθήσουν πολύ στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ και πρωτού κλείσουμε τη συζήτηση θέλουμε να ακούσουμε την Κομισιόν κυρία Μπάλτας. Σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που είμαι εδώ και χαίρομαι ακόμη για την ε, ενθουσιώδη συμμετοχή στη συζήτηση για τα σχέδια ψηφίσματος που αφορούν την κύρωση της απόφασης. 202 τροπολογίες, ε, εντυπωσιακός αριθμός που δείχνει το ενδιαφέρον. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχήν είναι αναφυσβήτητο ότι η Συμφωνία των Παρισίων ε, ήταν σημαντικό ορόσημο και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως ε, μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο πολυμερούς διακυβέρνησης. Βέβαια, πολύ γρήγορα υποχώρησε η εφορία και ο ενθουσιασμός. Εμείς ε, τον Μάρτιο ήδη δώσαμε την ανακοίνωση για το, τι μελγενέστε μετά το Παρίσι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης κύρωσης. Το το ίδιο αναφέρουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ότι χαιρετίζουν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισημαίνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ακυρώσει τη Συμφωνία των Παρισίων το συντομότερο δυνατό και εμπρόθεσμα προκειμένου να είναι συμβαλόμενα μέρη από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας αυτής. Όλα όσα έχουν μεσολαβήσει ε, από τότε δείχνουν την πλήρη δέσμευση και προσήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να διευκολύνει με κάθε ε, μέσο την την κύρωση και συνεργαζόμαστε με όλα τα θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Τώρα, για την ερώτηση Eckhout, για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και τις διαδικασίες τους. Υπάρχουν ε, συνταγματικές απαιτήσει ε, πρέπει να γίνουν σεβαστές ε, στα κράτη-μέλη. Και, και τα 28 κράτη-μέλη ελπίζουμε ότι μέχρι τα τέλη του 2016 θα τα καταφέρουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αναφέρεται και στις εξωτερικές μας παρουσιάσεις και στις συνομιλίες που θα έχουμε με και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις εθνικές διαδικασίες κύρωσης ε, για να προλάβουμε ε, να το καταφέρουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, με τις εθνικές εξελίξεις αυξάνεται η εσωτερική πίεση και περιμένουμε εν ώψη και του G20 και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα να αναγγείλουν ε, τις διαδικασίες που θα εφαρμόσουν για να κυρώσουν τη συμφωνία των ε, Παρισιών. Το ίδιο υποσχέθηκε ότι θα κάνει και η Βραζιλία πολύ γρήγορα και μάλιστα φαίνεται ότι ήδη 49 χώρες έχουν δηλώσει ότι θα είναι σε θέση να κυρώσουν την Συμφωνία των Παρισίων πριν τη, την ε, συνέλευση του Μαρακές, πριν την COP22. Οπότε πολύ πιθανόν να ξεπεράσουμε το 55% των παγκόσμιων εκλογών, ε, εκπομπών. Οπότε αυτή την άποψη θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να είμαστε και συνεπείς. Γιατί η κύρωση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Και είναι η απόδειξη της παγκόσμιας αποφασιστικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισιών. Αλλά η πράξη της κύρωσης ε, και οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς από μόνες τους δεν θα ε, πραγματοποιήσουν αυτή τη ρηξικέλευθη αλλαγή που περιμένουμε με την υλοποίηση των στόχων. Γιατί μόνο με εθνικές πολιτικές και μέτρα θα λάβει χώρα αυτή η αλλαγή. Και χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς πρωτοστατεί και με το νομοθετικό πακέτο και με τις δραστηριότητες ε, μεγάλης οικονομική εμβέλειας που προτείνουμε, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε το 40% άσχετα αν έχουμε κυρώσει τη συμφωνία και καταθέσει την κύρωση μέχρι τα τέλη του 2016. Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές στα, των μέσων του αιώνα, η Συμφωνία των Παρισίων καλεί ή προβλέπει την υποβολή τέτοιων στρατηγικών από τα μέλη μέχρι το 2020. Και μάλιστα εμείς έχουμε και τον οδικό χάρτη του 2050 που στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα και έχει πολύ ε, εξεζητημένα οικονομετρικά μοντέλα και βοηθάει τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν τις ενδιάμεσες στρατηγικές τους. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε και ε, την επιστήμη να ρημάσει και η IPCC μέχρι το 2018, μέχρι τον πρώτο διάλογο, ε, θα υποβάλει επιστημονική μελέτη σε με το σενάριο του 1,5 βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας, ε, γιατί ακόμη δεν υπάρχουν όλα τα ε, μοντέλα που χρειαζόμαστε. Οπότε περιμένουμε και τις επιστημονικές εξελίξεις για να αξιολογήσουμε το στόχο του 1,5%. Οπότε τέτοιου είδους ε, στρατηγικές το μέσο του αιώνα είναι σημαντικό στοιχείο και μέσω της πολιτικής για να μπορέσουν τα συμβαλόμενα μέρη να προετοιμαστούν και να καταρτήσουν και τα επενδυτικά τους ε, σχέδια για να διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και την Επιτροπή σας για την προσήλωσή σας σε μια ταχεία διαδικασία και νομίζω ότι πραγματικά είναι υποδειγματικός ο τρόπος ε, που διαχειρίζεται το θέμα και με την ανακοίνωση και εμείς πρωτοστατήσαμε και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί στις αποφάσεις του για να ακολουθήσει το παράδειγμα που βάλαμε. Και περιμένω με ανυπομονησία την έκβαση της ψηφοφορίας της 8 η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι η κύρωση της συμφωνίας, η έκθεση της κύρωσης συμφωνίας των Παρισίων η προθεσμία για τις τροπολογίες, μόνο στα αγγλικά όμως οι τροπολογίες, αύριο το πρωί στις 12 και θα ψηφίσουμε το τέλος, στο τέλος Σεπτεμβρίου για το ψήφισμα του Μαρακές. Μπορούμε να μεταφέρουμε την προθεσμία για τις χωριστές ψηφοφορίες και κατά τμήματα τη Δευτέρα 18 και θα ψηφίσουμε στις 8 Σεπτεμβρίου και θα γίνει η συνολομέρεια θα έρθει στις 8 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία. Θα ψηφίσουμε 8 και θα ψηφίσουμε την πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Δίνω τώρα το προεδρικό έδρανο στον Ζιλ Παρνιό. Enfin, chers collègues, donc euh, euh, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons et, et que je vais euh, pendant. Euh, Ευχαριστώ. Θα προεδρεύσω την επόμενη ώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και έχουμε τώρα στο επόμενο θέμα το σχέδιο δράσης κατά της λαθρεμπορίας αγρίων ειδών και θα δώσω το λόγο στην Κατερίνα Μπερντέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω με την έκθεσή μου, να δούμε τι είναι αυτή η εγκληματική δραστηριότητα ε, ε, με κύκλο εργασιών δισεκατομμύρια ευρώ από εγκληματικές ομάδες, συμμορίες που ασχολούνται και με ναρκωτικά, σωματεμπορία και ασχολούνται και με τα προϊόντα της άγριας ζωής όπως λέμε έχει υψηλή οικονομική απόδοση και χαμηλό ε, κίνδυνο σύλληψης και εντοπισμού. Είναι κάτι το οποίο αφορά την επιβίωση πάρα πολλών ανθρώπων στον πλανήτη. Είναι επίσης μια απειλή στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις τοπικές κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινότητες και στα οικοσυστήματα και καταλαβαίνετε ότι συνεισφέρει και στην απώλεια βιοπικιλότητας που δίνει ε, περιορισμένες δυνατότητες στον πλανήτη να συνεχίσει να λειτουργεί. Ε, δημιουργήθηκε με δική μου πρωτοβουλία πέρυσι η ομάδα Ευρωβουλευτές για την άγρια ζωή με πολλούς συναδέλφους Καφρόντε, Ζερόμ και τα λοιπά. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς για την διακομματική τους μορφή ενδιαφέροντος που μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Κάναμε συναντήσεις με ενδιαφερομένους, ξεκινήσαμε επαφές με το κοινό Ενθαρρύναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα πρόγραμμα δράσης και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον υπεύθυνο και το προσωπικό του, το οποίο προσπάθησε να κάνει κάτι γύρω από το θέμα αυτό. Ε, το σχέδιο αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ε, θα αντιμετωπιστεί είναι το πρόβλημα. Στην παράγραφο 9 της πρότασης τα κράτη-μέλη λέγεται ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα δράσης και να αναλάβουν ε, να κάνουν ενέργειες σε όλους τους σχετιζόμενους τομείς. Μπορούν να το κάνουν αυτό μόνο εφόσον υπάρχει διαφάνεια και σωστή αναφορά των προβλημάτων από όλα τα κράτη-μέλη. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μπροστά μας μια βολική, έτσι ευγενική ε, περιβαλλοντική πολιτική. Έχουμε θέματα εδώ ασφάλειας, ε, εμπορίου, δικαιοσύνης, ελέγχου συνόρων και αστυνόμευσης. Ε, καλύπτει πάρα πολλούς τομείς. Όλοι γνωρίζετε τι γίνεται με το ελεφαντόδοντο <clears throat> και ακούσαμε ότι μειώθηκαν κατά 20% οι, ε, οι πληθυσμοί των ελεφάντων στην Αφρική, κάτι το καταστροφικό. Αυτό αφορά όμως και τα φυτά ε, και τα λουλούδια και ακόμα όλα τα άλλα ζώα, τα αμφίβια, όλα όσα γίνονται αντικείμενο παράνομης εμπορικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Στην παράγραφο 23 βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες που φύγονται, όπως η βιομηχανία κατασκευής, παρασκευής τροφίμων, η μόδα και άλλες ε, βιομηχανικές ε, κυρίως δραστηριότητες. Εγώ στην έκθεσή μου λοιπόν λέω να δημιουργηθεί ένας συντονιστής καταπολέμησης των εγκληματικών δραστηριοτήτων εις βάρος της άγριας ζωής. Ε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έλεγα είναι καθρέφτης του προγράμματος που έχουμε δημιουργήσει για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Νομίζω ότι με τις διάφορες γενικές διευθύνσεις οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα και του τράφικινγκ και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, απαιτείται λοιπόν κάποιος ένα γραφείο συγκεκριμένα το οποίο να συντονίζει και να παρακολουθεί ε, πώς ε, ε, συλλέγονται οι πληροφορίες, πώς θα καταλήγουν όλες οι πληροφορίες σε ένα μέρος και νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο το οποίο δούλεψε καλά σε πάρα πολλές περιοχές και θα πρέπει να γίνει το ίδιο τώρα και εδώ. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την διαφθορά. Και να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση γι' αυτό. Είναι μια σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Αυτό έχει επιπτώσει όχι μονάχα στο διεθνές εμπόριο, αλλά και τη... υπάρχει εμπόριο όχι μόνο για άγρια ζώα από τρίτες χώρες, αλλά και από την Ευρώπη και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και πόροι <clears throat> στα σύνορα της Ευρώπης σημαίνει ότι μπορούν να έρχονται διάφορα άγρια ζώα χωρίς να το καταλαβαίνουν τελωνιακοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από τους τελωνιακούς, καλύτερη κατάρτιση για όλους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα αγαθά στον δρόμο τους στην Ευρώπη και η Ευρώπη δεν είναι μονάχα προορισμός αλλά είναι και περιοχή από την οποία προέρχονται αυτά τα άγρια είδη. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά και στην πηγή και στον προορισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ένα συστηματικό πλαίσιο για να μπορούμε να κατατίσουμε, να έχουμε αναφορές για τα θέματα αυτά, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και επίσης τα κρατημέλη ζητείτε να δημιουργήσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια Καλά είναι τα ευρωπαϊκά σχέδια, αλλά πρέπει να υπάρξουν και εθνικά σχέδια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και σε περιφερειακό και τοπικό. Όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα αν έχουμε ένα συντονιστή ο οποίο μπορεί να έρχεται σε επαφή με τα κράτη μέλη και να του ρωτάει τι κάνουν για να επιτύχουν το στόχο αυτό. Αν περάσουμε τώρα στο θέμα τη ε, αστυνόμευση, η Europol χρειάζεται ενίσχυση στο έργο του <clears throat> για το θέμα αυτό και η έκθεσή μου ζητά να υπάρξει μια ειδική μονάδα στην Europol για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο αγρίων ειδών. Χωρίς την πολιτική μας θέληση αυτό δεν θα γίνει. Το έγκλημα σε σχέση με τα άγρια είδη θα πρέπει να περιληφθεί μέσα στις απειλές από το οργανωμένο έγκλημα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο αυτή στιγμή και μας λέει η Europol δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν τεθεί στο σχέδιο δράσης για το σοβαρό έγκλημα. Αυτό πρέπει να προερθεί από τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Πρέπει η Ευρωπόλ να έχει λοιπόν τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εθνικές αρχές και πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά τους για σοβαρά εγκλήματα. Αυτό, αυτή η μορφή οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα με κοινή προσπάθεια και με, είναι απαραίτητο να υπάρξουν στρατηγικά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουν την αστυνόμευση. Και οι κυρώσεις τώρα. Πάμε τώρα στις ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται. Πρέπει να ενισχυθούν οι ποινές. Σε ορισμένε χώρες είναι πολύ ελαφρία η ποινή και η... δεν υπάρχει καμιά ποινή. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη προσπάθεια για να υπάρξουν ελάχιστες ποινές. Αυτό αναφέρεται στο σχέδιο δράση, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται πραγματικότητα και το Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει προστασία από τη Διεθνή Σύμβαση ΣΥΤΕΣ, αλλά μερικά ήδη δεν καλύπτονται από αυτό το πλαίσιο του ΣΑΙΤΕΣ. Πολλές χώρες έχουν καλές πολιτικές για τον τομέα του περιβάλλοντος, γιατί τα φυτά, τα ζώα προστατεύονται στις χώρες αυτές. Αλλά τα άγρια αυτά ήδη δεν έχουν καμία προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, οι Αμερικανοί έχουν το λεγόμενο νόμο Lacey και εμείς πρέπει να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Αν τα ζώα, αν τα φυτά έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προστατεύονται από το σύστημα CITES, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα τα κράτη-μέλη για να οδηγήσουν σε δίωξη τους λαθρεμπόρους τους. Πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν, κάτι αντίστοιχο με την νομοθεσία, με την πράξη λέηση στις ΗΠΑ, γιατί έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν το αγριοζωικό έγκλημα και μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Και επίσης η έκθεση τονίζει ότι το λαθρεμπόριο αυτό γίνεται πιο εύκολα επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Το εμπόριο για τα άγρια ήδη και φυτά, ζώα και φυτά, γίνεται πιο εύκολα στο διαδίκτυο. Αυτό τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να το δούμε αυτό και φυσικά αυτό βοηθάει και την έκπληση χρημάτων. Η συνεργασία λοιπόν στον χρηματοπιστωτικό τομέα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τα χρήματα αυτά, θα προστατεύσει καλύτερα τα άγρια είδη. Όπως και με οποιαδήποτε έκθεση μας περιορίζει ο χώρος και ο χρόνος, ο αριθμός των λέξεων και χαρακτήρων είναι εφιάλτης να περικόψουμε τον αριθμό των λέξεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ευζοία των ζώων που έχουν ως άγρια διασωθεί παρά τη λαθρεμπορία τους και θέλω εδώ να αναφερθώ σε αυτά που έχει κάνει το Βέλγιο, το οποίο έχει ένα θετικό κατάλογο για τα ζώα τα οποία <clears throat> επιτρέπεται να εισαχθούν, όχι μόνο να λέμε ε, τι δεν επιτρέπεται. έχουμε τη δήλωση του παλατιού του Buckingham για όλα αυτά τα θέματα και το να μπορέσουν όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί κλάδοι να ακολουθήσουν αυτή τη δήλωση είναι πολύ σημαντικό. Και τελικά τι είναι το άγριο. Τι είναι άγριο ζώο, άγριο φυτό. Είναι κάτι που το επεξεργάζεται το πρόγραμμα περιβάλλοντο των ΗΠΑ και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα σαφή ο οποίο να αναγνωρίζεται διεθνώ για το τι είναι άγριο και τι είναι ήμερο γιατί αλλιώς υπάρχει μια φαιά περιοχή. Πολλά λοιπόν είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στην έκθεσή μου και κάποια ακόμα στοιχεία θα τα προσθέσω ως τροπολογίες. Ευχαριστώ όμως τους ε, σκιώδεις συγητές, της ΜΚΟ, την Κομισιόν, τις εμπορικές οργανώσεις που έχουν βοηθήσει στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Έχουμε και άλλες συναντήσεις και σίγουρα θα υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες και εγώ θέλω τη συνεργασία σας όσο συζητάμε αυτές τις τροπολογίες και καταλήγουμε σε μια τελική έκθεση για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Merci, merci beaucoup, Σας ευχαριστούμε κυρία εισηγητρία για τις εξηγήσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στου σκιώδη εισηγητές. Η κυρία Πετήρ πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδη συγγήτρια του, κόμματος των Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπεάρντερ για την πολύ αξιόλογη της έκθεση και την προσπάθεια που κατέβαλε ε, για την προετοιμασία με επαφές με όλους τους αλλά και με συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές. Από διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, έμαθα πως κατά τη γνώμη τους το μείζον πρόβλημα σε σχέση με το λαθρεμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλεται στην ανεπάρκεια των ε, διοικητικών ικανοτήτων στα κράτη-μέλη. Ε, κυρίως ε, λόγω της έλλειψης ε, επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων, αλλά και λόγω της ανεπαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ανεπαρκούς διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μέλων. Γι' αυτό προτείνω να ενισχύσουμε τη διατύπωση για την ανάγκη κάλυψη αυτών των αδυναμιών. Θα σταθώ τώρα σε δύο παραγράφους που κατά τη γνώμη είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αναφέρθηκε σε αυτές και η κυρία Μπέρντερ η παράγραφος 19 αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστική παράγραφο, ικανοποιητική και δεν χρειάζεται να τη διαβρύνουμε περαιτέρω. Αυτή είναι η γνώμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. γιατί από τι πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε για την επίλυση τέτοιων θεμάτων, για παράδειγμα μέσω τη συμφωνία συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ, έχουμε καταλήξει σε πολύ καλά συμπεράσματα και τέτοιου είδου εμπειρίες θα πρέπει να τι χρησιμοποιήσουμε ω υποδείγματα των πρακτικών και στο μέλλον. Η παράγραφο 21 αφορά το διεθνέ εμπόριο ειδών. Χρήσιμη η αυτή, αλλά ο τρόπο με τον οποίο προτείνεται στην έκθεση αυτή δημιουργεί αμφιβολίες για την ασφάλεια δικαίου φυσικών και νομικών προσώπων που ασχολούνται με το εμπόριο εξωτικών ειδών. Για παράδειγμα, η απέτηση παροχής πληροφοριών για το καθεστώς των ζώων στις χώρες προέλευσης. Είναι κάπως αφιλεγόμενο. Γιατί αυτό το σκοπό εξυπηρετούν κατάλογοι όπως αυτή της σύμβασης σε σάιτες. Ε, να έχουμε δηλαδή ενιαίους καταλόγους προστατευμένων ειδών που να εφαρμόζονται πάντως στον κόσμο. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, δημιουργούνται κάποια, κάποιοι προβληματισμοί ασφάλειας δικαίου που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η κυρία Μπεάρντερ επικεντρώθηκε στο ουσιώδες, την αναχέτηση δηλαδή του λαθρεμπορίου άγριας χλωρίδας και πανίδας και ελπίζω αυτή η έκθεση να παραμείνει ε, συνοπτική, μεστή και σημαντική και να μην επεκταθεί σε περαιτέρω άχρηστα σημεία. Θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου προς την εισηγήτρια. Σας ευχαριστούμε κυρία Πετήρ, την κυρία Μελχιόρ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Καταρίνα Μπέρντερ, για την πολύ καλή ε, εξισορροπημένη και φιλόδοξη έκθεση της. Είμαι πεπισμένη ότι ανεξάρτητα από πολιτικές ομάδες θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι σε μια έκθεση η οποία θα δώσει τις σωστές κατευθύνσεις για να αντιμετωπίσουμε το παράνομο εμπόριο ζωικών και φυτικών ειδών. Η κυρία Μπέρτερ έχει αναφερθεί σε πάρα πολλές σημεία. Εγώ θα σταθώ μόνο σε τρία τα αυτά τα σημεία. Πιστεύω <clears throat> ότι χωρίς την συμμετοχή και την θέληση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μια τέτοια ενέργεια και θα αποτύχει και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου έχει χαιρετιστεί το σχέδιο δράσης, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία συγκεκριμένη υπόσχεση σε ό,τι αφορά την διάθεση πόρων ή προσωπικού για την υλοποίηση αυτού του σχέδιου. Αυτό είναι όμως σαφές, όπως είπε και η κυρία Μπέρντερ, ώστε να μπορέσει να αναχαιρετιστεί το, ε, το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών στην γερμανική Bundestag, στη χώρα μου. Υπήρξε τον Ιούλιο μια απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού για να αντιμετωπιστεί αυτή η προβληματική <clears throat> και ελπίζω ότι και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο θέμα αυτό και αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα για την πρόοδο. Υποστηρίζω λοιπόν απόλυτα, όπως είπε και η κυρία Μπέρντερ, ότι οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να αντανακλούν το περιεχόμενο του νόμου Λέιση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία ειδών και ζώων που δεν θα πρέπει να εισάγονται στις χώρες μας εάν προστατεύονται στις χώρες τους αλλά δεν υπάρχει κάποια διεθνής προστασία για τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια πραγματική εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των αγρίων ειδών και ότι θα μπορέσει να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή και αστυνόμευση στα κράτη-μέλη. Επειδή τώρα έχουμε μία συζήτηση πολλές φορές για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία έχουν προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει στις συμφωνίες αυτές να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η προστασία των αγρίων, ζωικών και φυτικών ειδών. Επομένως, αυτό αφορά και τη συμφωνία με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε κάποτε να τη ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει μέσω των εμπορικών αυτών συμφωνιών να κάνουμε τα απαραίτητα για να υπάρξει η προστασία των ε, ειδών αυτών, των αγρίων αυτών ειδών και ελπίζω ότι στο μέλλον θα παίξει κάποιο μεγαλύτερο ρόλο αυτή η προστασία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία εισηγήτρια και είμαι πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ωραία έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ντέμες Μάκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο μας εδώ και πάρα πολύ καιρό υποστηρίζει το να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της λαθρεμπορίας αγρίων ζωικών και φυτικών ειδών. Αυτού του είδους το εμπόριο είναι θανατηφόρο για την βιοπικιλότητα και πάρα πολλά από αυτά τα ζωικά είδη θανατώνονται. Ήδη από το 2013 είναι πάνω από 20.000 ελέφαντες από τότε μέχρι σήμερα που έχουν θανατωθεί. Αλλά υπάρχουν και άλλες ολέθριες συνέπειες του εμπορίου αυτού. Είναι εκατομμύρια ε, ευρώ τα οποία περνάνε με τον τρόπο αυτό στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων και τρομοκρατικών οργανώσεων που μπορούν να συνεχίσουν τις δράσεις τους. Τρία τέταρτα του ε, παράνομου εμπορίου ε, του γίνεται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Επομένως, η δράση μας είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε και την προστασία των αγρίων ειδών, αλλά και την ασφάλειά μας. Όπως είπε λοιπόν και η συγγήτρια πρέπει να κάνουμε πολλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξετάσουμε καλύτερα την ε, ε, προέλευση αυτών των ειδών ή τη διέλευσή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράση το οποίο δημιούργησε η Κομισιόν τον ε, Φεβρουάριο έχει ένα θετικό χαρακτήρα. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί και η αποτελεσματική του εφαρμογή σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα να γίνουν πραγματικότητα και όπως είπε και η συγγήτρια, είναι πολύ καλό να αναφερθούν οι βέλτιστες πρακτικές μεταξύ άλλων και στη δική μου χώρα. Εγώ χαίρομαι λοιπόν που θα μπορέσει να γίνει αυτή η προσπάθεια για την καλύτερη εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα η κυρία Μπέρντερ με την έκθεσή της και έχει την εστίαση αυτή. Έχουμε μια σωστή έκθεση και μια φιλόδοξη έκθεση. Έχω καταθέσει μια σειρά, μια περιορισμένη ομάδα τροπολογιών και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπέρντερ για την προδραστική και επικοδομητική της στάση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου με το περιεχόμενο της έκθεσης ε, της κυρίας Μπεάρνταρ. Και διαπίστωσα με χαρά ότι αναφέρεται η ανάγκη να τροποποιηθεί το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο για να απαγορευτεί η πώληση προστατευμένων ειδών στις χώρες προέλευσής τους και που παράνομα ε, έγιναν αντικείμενο κυνηγιού και κατόπιν ε, μεταφοράς για εμπορία σε άλλη χώρα. Και όπως είπε, καλό θα ήταν να μιμηθούμε το παράδειγμα των Αμερικανών, την νομοθετική πράξη λέει, Συμφωνώ μαζί της. Επίσης, είχαμε και την σχετική εκθέση του Κοινοβουλίου για το οργανωμένο έγκλημα κατά της Άγρες Πανίδας. Ε, έχουμε μελέτες των κυβερνητικών οργανώσεων και είναι σημαντικό και το, το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου αυτού να αντανακλά όλες αυτές τις προεργασίες που έχουν γίνει. Επίσης θα πρέπει να, κατα, να καταπολεμήσουμε την ε, γενικευμένη διαφθορά που διέπει αυτό το λαθρεμπόριο άγριας ε, φλόριδας και πανίδας και να το αντιμετωπίσουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Γιατί ε, ένα σοβαρό οργανωμένο έγκλημα μόνο από μια σοβαρά οργανωμένη προσπάθεια και έναν σοβαρό μηχανισμό επιβολής και προστήμων ποινών θα αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ισχυρό μηχανισμό για να εξασφαλίσουμε την επιβολή και να ε, βρούμε τους απαραίτητους πόρους ε, για να χρηματοδοτήσουμε τα διαδοχικά στάδια που προβλέπει το σχέδιο δράσης. Και επίσης ε, να φροντίσουμε για τα ζώα που έχουν κατασχεθεί και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία και να τη χρηματοδοτήσουμε για να μην μένουν α, στο, στη μοίρα τους αυτά τα ζώα. Επίσης, να ενισχύσουμε την προστασία και την συνεργασία μεταξύ των μονάδων προστασίας της Άγρια Πανίδας. Σε ό,τι αφορά τα θέματα του εμπορίου, ε, θα ήθελα οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε να περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εφαρμόσιμες διατάξεις για την εφόρο ανάπτυξη. Γιατί έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι η συμπερίληψη ε, τέτοιων θεμάτων σε εμπορικέ ε, ε, συμφωνίες είναι μόνο για καλοπιστικούς λόγους. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να εφαρμόζω τέτοιες διατάξεις για την προστασία των ζώων και να υπάρχουν και συνέπειες ε, για αυτούς που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τέτοιες διατάξεις. Αυτά και είναι πολύ ε, ελπιδοφόρα η πρόταση. Θα την ε, επεξεργαστούμε περαιτέρω με τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριο Σαφρόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια κατανοώ γιατί είναι περιορισμένη σε μέγεθος η έκθεση, αλλά είναι σαφής. Καλύπτει νομίζω όλη τη θεματολογία του προβλήματος αυτού. Ένα πρόβλημα το οποίο ε, έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να αντιμετωπιστεί επιγόντως. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα στα πλαίσια των τροπολογιών. Ένα σημαντικό θέμα είναι το 5 για την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη μείωση στην αγορά αυτών των προϊόντων. Είναι σημαντικό εδώ το θέμα να μιλήσουμε για ελέγχους, για οδηγίες, για κανονισμούς. Αλλά σημασία έχει να αλλάξουμε, θα έλεγα, ε, την ε, κουλτούρα αυτών οι οποίοι καταναλώνουν τέτοιου είδους προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ένα θέμα το οποίο είναι όλο ένα πιο περιφερειακό αν θέλετε, το θέμα των μη θελημένων συμπεριφορών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν και έρχονται πίσω με ζώα ή με τμήματα ζώων που δεν γνωρίζουν ότι απαγορεύεται να τα θανατώνουν και να τα εισάχουν. Πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν, να λέμε ότι αν πηγαίνετε σε αυτή τη χώρα να δείτε ότι θα βρείτε σουβενίρ αναμνηστικά ε, κάποιου τύπου, αλλά να ξέρετε ότι απαγορεύεται να τα αγοράσετε και να τα εισάγετε στη χώρα σας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια συμπληρωματική εκστρατεία ενημέρωση σε σχέση με αυτή που προτείνει η συγγήτρια, αλλά πρέπει να την υπογραμμίσουμε. Ε, είναι καλή πρόταση για να δημιουργηθεί επίσης και ένας, διεθνή, ένας Ευρωπαίος συντονιστής για την ε, καταπολέμηση της δραστηριότητας αυτής. Θα πρέπει η προσπάθεια όμως να γίνει κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών. Πολλές φορές έχουμε σωστές στρατηγικές, σωστές οδηγίες, οι οποίες γενικά ξεκινούν με σωστό τρόπο, αλλά φοβάμαι ότι μετά χάνονται κάπου στην μετάφραση. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη να παρεμβαίνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μια άλλη ανησυχία μου είναι η έλλειψη ισορροπίας που θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χώρες. Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και διαθέτουν πόρους και προσωπικό για να αντιμετωπιστεί, πολλές φορές δημιουργεί ε, προβλήματα ε, διαφορών ανάμεσα σε χώρες και αυτό δημιουργεί νέους διαδρόμους ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ε, ασκούν παράνομες δραστηριότητες στις χώρες όπου γνωρίζουν ότι το κράτος παρεμβαίνει όλο και λιγότερο. Απαιτείται λοιπόν αυτή τη στιγμή μια θα έλεγα μορφή συντονισμού έτσι ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικά τύχη εναντίον αυτής της δραστηριότητας. Στο σημείο 10 καλούνται τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα έτσι ώστε οι υποδομές αυτές να έχουν τους απαραίτητους διαθέσιμους πόρους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσει κάποια χρήματα για αυτήν την ε, ε, δραστηριότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες αντίστοιχες δραστηριότητες. Αναφέρεται το θέμα ε, των πόρων, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν ταμεία από τα οποία θα μπορούσε να προέλθει, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, αν μπορεί να υπάρξει εκεί μια θέση συγκεκριμένη για αυτού του είδους ε, την μάχη η οποία θα πρέπει να δοθεί. Σημαντική και η αναφορά στο σημείο 9, όπου καλούνται τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα εθνικής δράσης, Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ε, επιλέξουμε τη σωστή μέθοδο και τον σωστό τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν δράση από πλευράς των κρατών μελών ή αν υπάρξει έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά τα οποία θα κάνουν τα κράτη-μέλη, τότε έχει σημασία να δούμε αυτό που λέει το σημείο 5 της έκθεσης, ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει σε αιτήσια βάση να παίρνουν γραπτές, να λαμβάνουν γραπτές εκθέσεις από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της στρατηγικής των κρατών μελών. Έχει σημασία να παρακολουθείτε από κοντά το πώς εφαρμόζεται αυτή η προσπάθεια από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αποφύγουμε να βρεθούμε πέντε χρόνια μετά από την υιοθέτηση για την βιοπικιλότητα στην έκπληξη που θα λέει ότι δεν πετύχαμε τους στόχους. Και όλα αυτά όπως είπα στα πλαίσια μιας στρατηγικής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι αποτελεσματική και θα έρθει και η έκθεση της δικής μας Επιτροπής, μια πολύ θετική έκθεση που θα μας βοηθήσει να συντονιστούμε ακόμα καλύτερα. Ο κύριος Γκερμπράντ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Κάθριν Μπάρντερ για την εξαιρετική της έκθεση και για το ότι διάλεξε αυτό το θέμα και το ανέπτυξε με τόσο προσιλωμένο τρόπο. Όταν πριν από μερικά χρόνια αρχίσαμε να ε, ασχολούμαστε με το θέμα και εγώ υπέβαλα το δικό μου σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, τραβήξω την προσοχή σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, οι αρχικέ αντιδράσει δεν ήταν και πολύ ελπιδοφόρε. αλλά τελικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστερνίστηκε αυτή την πρόταση και κατέθεσε τελικά ένα σημαντικό σχέδιο δράσης ε, και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πυγμή που έδειξε. Και εμείς ε, είχαμε ζητήσει έντονα κάποια πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε προσήλωση και έρχομαι στο τρίτο θεσμικό όργανο, το Συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Γιατί αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί εκεί λαμβάνει η χώρα η εφαρμογή, η εκτέλεση, η αστυνόμευση. Εκεί οργανώνεται σε εθνικό επίπεδο. Και θα ήθελα να τονίσω και πάλι πόσο βαθιά με απογοήτευσαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου επί Ολλανδικής Προεδρίας και τα σχόλια για το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν εξετάσουμε όλη τη δέσμη δράσεων του σχεδίου δράση, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλες εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και η δέσμευση δυστυχώ των κρατών μελών ε, παρά είναι ε, ασθενή ε, και δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Και πρόσφατα έγινε σαφές πόσο σημαντικό είναι το θέμα γιατί η τελευταία μελέτη για τους μελέτες στην Αφρική δείχνει ότι το 1 τρίτο του συνόλου των ελεφάντων θανατώθηκαν μεταξύ 2007 και 2014. 1.400 ε, ελέφαντες έχουν σφαγιαστεί από ε, αχρίους και έχουμε ελάχιστους ελέφαντες που μας έχουν απομείνει και αυτό δεν αφορά μόνο τους ελέφαντες αλλά και άλλα ζώα στον κόσμο, στη φύση. Τεράστιο λοιπόν το πρόβλημα, οξύτατο και με απογοητεύει ιδιαίτερος η στάση των κρατών μελών. Για μένα το σημαντικότερο σημείο της έκθεσης είναι η έκκληση για άσκηση πίεση στα κράτη-μέλη για να κάνουν το καθήκον τους, για να διασώσουμε την άγρια χλωρίδα και πανίδα στον κόσμο. Και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επαναλαμβάνω ιδιαίτερω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Κάθριν Μπεάρντερ. Και πιστεύω ότι μπορούμε με συλλογική προσπάθεια να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ήδη αξιόλογη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Γκερμπράντε. Η κυρία Κάντεμπαχ τώρα. Ja, ein herzliches Dankeschön. Auch ich möchte mich bei Catherine bedanken. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κάτριν Μπέρντερ και όλους τους συναδελφούς οι οποίοι προελάλησαν εμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι και στα κράτη-μέλη μας ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μονάχα η προστασία της βιοποικιλότητας δεν έχει να κάνει μονάχα με, την, ε, με τις δηλώσεις αυτά που γράφει κανείς σε μια αφίσα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε τα απαραίτητα για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο με τα άγρια ζωικά είδη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σημαντική υποστήριξη ούτε σε πολιτικό επίπεδο ούτε και από την κοινή γνώμη. Δεν υπάρχει απαραίτητη συνειδητοποίηση. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να το φέρει κανείς στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο περιορίζεται η βιοπικελότητα το εμπόριο αυτό ε, αγριονιδών. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν όλοι να κάνουν το αντίθετο, να κάνουν μειώσεις στο προσωπικό και στα μέσα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και είναι σαφές ότι σε πολλά κράτη-μέλη οι υπάρχουσες οδηγίες και κανονισμοί εφαρμόζονται με πολύ εμβαλωματικό και περιορισμένο τρόπο και δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και πρέπει να θέσουμε μια έμφαση στην καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες μας. Θα πρέπει να καταλάβουν την ανάγκη για την προστασία της βιοπικελότητας και της άγριας ζωής και να καταλάβουν ότι πρέπει αυτές οι ενέργειες να έχουν τον απαραίτητο προϋπολογισμό και επομένως <clears throat> ότι η εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπομειστεί και με το έργο του ελέγχου στα θέματα αυτά. Μόνο αν ξέρουν οι πολίτες μας την προβληματική και κατανοούν τι γίνεται, είναι σε θέση να υποστηρίξουν μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση και μια μεγαλύτερη στελέχωση με προσωπικό. Επομένως, από την πλευρά της Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για να υπάρξει πρόθεση αυτού του θέματος. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η απαραίτητη θέση σε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή ημερήσια διάταξη και σας λέω και πάλι είναι απαραίτητο να ασκήσουμε την πίεση που χρειάζεται στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος, κυρία Καλντέμπαχ. Ο... Κυρία Μέιερ για την Κομισιόν έχει το λόγο. και κύριοι, καταρχάς θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε και σα σαν Επιτροπή και την εισηγήτριά σα, όπως και όλους όσους ε, έχουν ε, προσφέρει τις δικές τους προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους ε, λαθρεμπορία ε, πολιτήμων ειδών που προέρχονται από ζώα ή επίσης ε, και καταπολεμήσουμε τις ενέργειες της βάρος της άγριας ζωής. Η προσπάθεια που γίνεται γίνεται σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπηρεσίες των διαφόρων Υπουργείων των κρατών μελών. Μόνο ο σωστό συντονισμό θα μα επιτρέψει τη σωστή καταπολέμηση αυτή τη εγκληματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες νέες προτάσεις, πέραν αυτών τις οποίες προτείναμε τον μήνα Φεβρουάριο. Γνωρίζετε ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με την απειλή εις βάρος των αγριών ζώων παραμένουν οι Ολλανδοί ε, τελωνιακοί ε, δύο τόνους προϊόντα κατέσχεσαν πρόσφατα, είτε κοράλια, είτε κρανία πυθίκων και μάλιστα είχαν βρει μαζί με τα ίδια αυτά, τα, παράνομα, τα παρανόμως σε βασί περιπτώσει η λεγέντα, είχαν βρει επίσης και 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας. Συνεπώς λοιπόν το Συμβούλιο ε, έχει ενισχύσει την προσπάθεια η οποία γίνεται και οι προσπάθειες αυτές θα συνεχίσουν να γίνονται και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Europol και σε επίπεδο Eurojust. Έτσι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε από κοντά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, ξεκινώντας α, στις αρχές του 2017 και ε, συνεχίζοντας και με μια διαφανή έκθεση για τα βήματα προόδου τα οποία έχουν ήδη επιτελεστεί. Η διεθνή συνεργασία είναι θα έλεγα κάτι το καθοριστικό ε, η διάσκεψη των συμμετεχόντων στην ε, σύμβαση ΣΥΤΕΣ ε, θα συνεδριάσει σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συνεχίσει τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει και στον τομέα των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών για να χρησιμοποιήσουμε το εμπορικό βάρος της Ένωσης και να επηρεάσουμε θετικά την καταπολέμηση αυτής της δραστηριότητας. Πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση για τα προϊόντα αυτά σε ασιατικές κυρίως χώρες και ενισχύουμε όλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει άλλο ένα σημείο επιπλέον το οποίο θα ήθελα να σημειώσω που συνδέεται με την παράγραφο 21 της έκθεσης για την προστασία από πλευράς τρίτων χωρών ορισμένων ειδών. Κάτι το οποίο ξεπερνά την προστασία την οποία παρέχει οι ΣΥΤΕΣ μέχρι τώρα και την ανάγκη να υπάρξει θα έλεγα ένας ευρωπαϊκός νόμος ο οποίος θα μπορέσει να λειτουργήσει σε συγχρονία με το Lacey Act, το νόμο Lacey στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τις χώρες οι οποίες θέλουν να, να δημιουργήσουν ένα μητρό μέσω της σύντες των ειδών τα οποία απειλούνται. Εμείς ε, το κάνουμε συχνά αυτό. Ε, ερχόμαστε σε επαφή με τρίτες χώρες που εξηγούν το πρόβλημα το οποίο έχουν ε, για τις απειλές, με τις απειλές εις βάρος των ειδών και βοηθούμε τις χώρες αυτές και σε επίπεδο επιστημονικό και σε επίπεδο πολιτικό να προετοιμάσουν ε, την ε, ε, προσπάθειά τους καταλογοποιώντας κατά κάποιο τρόπο τα παραρτήματα τα ίδια αυτά. Και έτσι η προστασία δεν είναι μια προστασία αποκλειστικά εις βάρος της ευρωπαϊκής, αποκλειστικά σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι οι ΣΥΤΕΣ μπορεί να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά και είναι και μια διαδικασία λιγότερο, περισσότερο ευέλικτη σε επίπεδο διοικητικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προσπάθειες τις οποίες έχετε μέχρι τώρα κάνει και θα παρακολουθήσουμε από κοντά την έκθεση αυτή όταν γίνει δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Να σας διευκρινίσω. Α, συγγνώμη. Η συγκεκριά κυρία Μπέρντερ, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Είναι πολύ ενθαρρυντικό με το που ε, ανοίγουμε το μικρόφωνο αρχίζουν να χτυπάνε και το τηλέφωνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, με εγκαρδιώνει ιδιαίτερα η θερμή υποστήριξη των συναδέλφων για την έκθεσή μου. Και επίσης είστε υπέρ και των συγκεκριμένων δράσεων, της ανάγκης διαφάνεια και της έκκληση προ τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση και να συνεργαστούν μεταξύ τους γιατί κάθε νέα πρωτοβουλία απαιτεί χρήματα και είναι δύσκολη η ανέβρεση χρηματοδότησης και χαίρομαι που συμφώνησαν και με αυτό οι συνάδελφοι. Γιατί και στην δική μου χώρα όταν ε, ψάχνουμε πού θα κάνουμε τις περικοπές ε, το μεγαλύτερο θύμα είναι το περιβάλλον και το βλέπουμε εδώ και στην Επιτροπή πως το περιβάλλον είναι φτωχό συγγενής όταν θέλουμε να κάνουμε οικονομίες. Και φυσικά χρειαζόμαστε πόρους ε, και όλα αυτά κοστίζουν, έχουν ένα τίμημα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες από τα κράτη-μέλη και να αναζητήσουν πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, ε, ε, ιδιαίτερα στην Αφρική, το οργανωμένο έγκλημα κατά της άγριας ζωής ε, είναι εντυπωσιακό και οδηγεί και στο ρήγμα, σε ρήγματα, σε ρήξεις μεταξύ των κοινωνιών με συμμετοχή και του στρατού και όλοι έχει ε, συνέπειες και στη μετανάστευση. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα να εξετάζουμε πρώτα τα αίτια του, τη ρίζα του προβλήματος. Είναι τεράστιες συνέπειες και στο, στις κλιματικές αλλαγές, στο περιβάλλον, όλα είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να εγγύψουν στο θέμα και να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ για την στήριξη που δώσατε στις, στις εκστρατείες που πρότεινα αφύπνισης, γιατί μερικές φορές ο τελευταίος που γνωρίζει τα πράγματα είναι ο καταναλωτής. Θα πρέπει να τον ενημερώσουμε ε, ώστε όταν αγοράζει μια χελώνα είτε όταν τρώει ποδαράκια παλεπού ή να ξέρει ε, ότι αυτά μπορούν να ανήκουν σε προστατευμένα είδη. Οπότε και δεν θα πρέπει να κάνουμε εύκολη τη ζωή στους ε, εγκληματίες. Επίσης είχαμε αυτή τη Lacey Act, αυτό το νομοθέτημα των ε, Αμερικανών, που θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε, να μιμηθούμε αυτές τι προτάσεις και να συμπεριλάβουμε στι εμπορικές μα συμφωνίε. Και οι σάιτες, οι συμφωνίες σάιτες είναι πολύ καλή παγκοσμίω για τα απειλόμενα είδη, αλλά είναι πολύ ε, βραδικίνητη διαδικασία γιατί απαιτούνται συνεδριάσεις των ε, ε, επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων, κάτι που καθυστερεί την όλη διαδικασία. Και Μερικέ χώρε έχουν κάποια ζώα που είναι σημαντικά για το οικοσύστημά του και απειλούν τη χρήση προστασία στη, χώρα αυτή, αλλά δεν προστατεύονται παγκοσμίω. Αλλά δεν εμπίπτουν αυτά τα ζώα στην ε, Συμφωνία Σάιτε. Αλλά για τη συγκεκριμένη χώρα υπάρχει ε, νομοθεσία που προστατεύει το συγκεκριμένο φυτό και το καθεξής. Οπότε, σε περίπτωση που γίνεται εξαγωγή αυτού του προστατευμένου είδου, ε, ε, ζημιώνεται η συγκεκριμένη χώρα όχι ο παγκόσμιος πληθυσμός και σε τέτοιες περιπτώσεις η πρόοδος είναι αρκετά πιο αργή. Αν λοιπόν πούμε ότι σε περίπτωση που είναι παράνομη εξαγωγή σε μια χώρα θα σεβαστούμε αυτή την απαγόρευση και θα σταματήσουμε να εισάγουμε αυτό το αντικείμενο, το ζώο ή το φυτό. Και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι κατά του πολλαπλασιασμού των νομοθετικών προτάσεων, αλλά μερικές φορές χρειάζονται. Και αν εξασφαλίσουμε προστασία της άγριας χλωρίδα και πανίδα στον κόσμο και στηρίξουμε τις χώρες στην περιβαλλοντική του πολιτική, ε, θα είναι ευάρεστο. Και ευχαριστώ τους και ηγετές και τους συναδέλφου γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι κατεπήγον. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να επιληφθούμε μετά από μία πενταετία. Οπότε, όσοι ασχολείστε με το θέμα αυτό, όποιος ευρωβουλευτής ε, ε, έχει κάποιον υπουργό περιβάλλοντος στη χώρα που δεν έχει καταλάβει το μήνυμα, ε, πάτε προτείνει του μια επίσκεψη ή αυτόν ή την οικογένεια του, τα παιδιά του, για να καταλάβουν την απειλή που ισχύει για την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, και με την έκθεσή μα να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία τη με τα κράτη-μέλη, αλλά και μεμονωμένα μονομένα ως πολιτικοί μπορούμε να έχουμε επαφέ με εθνικού πολιτικού ε, για να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να ληφθούν κατεπηγόντω δράσει. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά ε, το πρόβλημα της τεράστια καταχρήση που γίνονται ει βάρο του περιβάλλοντο. Ευχαριστώ πολύ κυρία και το σύνολο αυτών που έλαβαν χώρα, έλαβαν μέρος στη συζήτηση για την ποιότητα των ε, ε παρεμβάσεών τους. Το χρονοδιάγραμμα μας για αυτό το κείμενο τώρα έχει ως εξής. Οι τροπολογίες μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 13 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια. Θα πάμε τον Νοέμβριο. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας και θα ξαναβρεθούμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Χένβη στις 8 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Αλλά θα έχουμε και μια έκτακτη συνεδρία στις 12 Σεπτεμβρίου στο Στασβούργο. Καλή όρεξη.